So, good morning everybody. Uh, I'm... Καλή σας μέρα. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας, λέει η Πρόεδρος, αλλά δεν έχουμε εικόνα. Χαίρομαι που σας βλέπω ακόμα και εξ αποστάσεως. Πρέπει όμως να δουλεύουμε 100% εξ αποστάσεως για να αποφύγουμε στο ελάχιστο τις ε, επαφές. Έγκριση του σχεδίου μερίσιας διάταξης πρώτα. Εγκρίνεται αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν βλέπω στην οθόνη μου κανέναν να ζητάει το λόγο, να έχει αντίρρηση, οπότε εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Επίσης, τα πρακτικά των δύο τελευταίων συνεδριάσεων. αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. 16 Οκτωβρίου πρώτα απ' όλα και 29 Οκτωβρίου. Υπάρχουν, δεν βλέπω να υπάρχουν ε, αντιρρήσεις για αυτά. Οπότε περνάμε στο τρίτο σημείο, μετά τα πρακτικά, το οποίο θεωρούνται εγκεκριμένα. Και τώρα σήμερα θα έχουμε, πιστεύω, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Τροφίμων Υπάρχουν πολλές ανησυχίες όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε για την πρόσφατη εντολή τους όσον αφορά αυτό το θέμα. Και πριν ξεκινήσουμε θέλω να σας δώσω κάποιες οδηγίες, να σας υπενθυμίσω κάποια πράγματα για αυτές τις εξαποστάσεως συναντήσεις. Ξέρετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την διερμηνία. Σήμερα έχουμε διερμηνία στα γαλλικά, στα γερμανικά, στα ιταλικά, στα ολλανδικά, στα αγγλικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα πορτογαλικά, τα σλοβενικά, τα ουγγρικά, τα σλοβακικά και τα ρουμανικά. Σας υπενθυμίζω επίσης, εφόσον παίρνετε το λόγο, φροντίστε να υπάρχει εικόνα και να χρησιμοποιείτε και ακουστικά όσο μπορείτε, γιατί έτσι ο ήχος σου βγαίνει καλύτερα αν δεν υπάρχει εικόνα, δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε και την μετάφραση, τη διερμηνία. Και μην ξεχνάτε, αυτή είναι η φράση της χρονιάς, πατάτε το κουμπί ομιλία για να πάρετε το λόγο. Περνάμε λοιπόν τώρα στην ουσία τη σημερινή μα συνεδρίαση. Πρόκειται για την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη διάρκεια τη μεταφορά. Και θα την παρουσίαση του Νίκολαου Κρίτ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλεια Τροφίμων. Ο ίδιο είναι κτηνίατρο και χαίρομαι επίση που και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα σήμερα με τον Κρίστιαν Τζούλιουσον από την Γενική Διεύθυνση Υγείας. Οπότε μαζί με τον ε, κύριο Κρίτ θα απαντήσουν στι ερωτήσει μα. Πρώτο, ο κύριο Κρίτ θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση όσον αφορά την εντολή τη ΕΦΣΑ που έλαβε από την Επιτροπή τον Ιούνιο για να ετοιμάσει γνωμοδότηση όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την μεταφορά του. Έχει μόλις ξεκινήσει το έργο τους και έχουν μέχρι τον Ιούνιο του 2022 για να ετοιμάσουν την γνωμοδότησή τους. Έχουν περισσότερο χρόνο από εμά δηλαδή. Αλλά ο κύριο Κρίτ έχει ήδη ετοιμάσει διάφορε εκθέσει όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων και θα μας μιλήσει για την ε, γνώση που ήδη υπάρχει στην ΕΦΣΑ όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ε, ζώων. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι εδώ επίσης για να απαντήσει στις ερωτήσεις μας. Ω ήθεστε λοιπόν, ξεκινάμε με την παρουσίαση του κύριου Κρίτς και μετά θα έχουμε χρόνο για ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα λοιπόν, καλωσορίζουμε εδώ και δίνω το λόγο στον κύριο Κρίτς για 15 λεπτά για να μας κάνει την παρουσίαση αυτή. Ευχαριστώ πολύ. Morning. Good to see you. Καλημέρα και καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ε, Πρόεδρε και αγαπητά μέλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ελπίζω να μ' ακούτε καλά θα ήθελα καταρχάς να σας συστηθώ σύντομα και να σας ευχαριστήσω ήδη για την δική σας εισαγωγή. Λέγομαι Νίκολαος Κρίτς και είμαι τμήματάρχης ε, για ε, την υγεία των ζώων, την ευημερία των ζώων και την υγεία των φυτών στην ΕΦΣΑ. Την τελευταία φορά που είχα το προνόμιο να έρθω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν το Φλεβάρι. Άλλη καιρή τότε, με αυτό παρουσία στην Επιτροπή Γεωργίας για να παρουσιάσω ε, την επιστημονική μας γνωμοδότηση ε, για τη σφαγή κονίκλων και την κονικλοτροφία επίσης. Ε, το Κοινοβούλιο μας ζήτησε να γνωμοδοτήσουμε τότε και το σημαντικότερο που θέλω να πω και να τονίσω είναι ότι έχω πάρα πολύ αφοσιωμένους νέους επιστήμονες και διοικητικούς υπαλλήλους που είναι πρόθυμοι να συνεισφέρουν θετικά στις συζητήσεις αυτές και να συνεργάζονται ιδιαίτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το έχουμε κάνει ήδη σε δύο άλλους τομείς στην ευημερία των ζώων και για την μελισσοκομεία και ε, την υγεία των μελισσών. Αυτό δεν είναι πάρα πολύ κοινό, αλλά είναι πάρα πολύ ευπρόσδεκτο, όπως σας είπα το Φεβρουάριο. Και είναι κάτι σίγουρα το οποίο υπερβαίνει την κανονική δουλειά που κάνουμε με τα κράτη-μέλη και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ό,τι αφορά την ευημερία των ζώων στη μεταφορά, που είναι η δική σας Επιτροπή ε, και το δικό σας θέμα, να σας εξηγήσω λίγο τι κάνει η ΕΦΣΑ για την υγεία των ζώων και την ευημερία τους και μετά θα επικεντρωθούμε, όπως είπατε και εσείς, ε, στις εντολές ε, που έχουμε ειδικά λάβει για τη μεταφορά των ζώων και να συζητήσουμε λίγο περισσότερο το ότι μελιγενέστε λιγενέστε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, να μας βοηθήσετε κι εσείς στην εργασία μας και να συμμετέχετε περισσότερο σε αυτή. Το σημαντικό ε, ε, είναι να πούμε τι είναι η και τι δεν είναι. Δημιουργήθηκε, συστήθηκε το 2002 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Τροφίμων και ήδη από τότε οι νομοθέτες ε, ε, και οι βουλευτές είχαν την πρόνοια να προσθέσουν δύο πάνελ για την υγεία και την ευημερία των ζώων το ένα και το 2006 το πάνελ για την υγεία των φυτών ε, για να μην μιλάμε μόνο αμυγός για την ασφάλεια των τροφίμων, αλλά και για επιπλέον μέτρα που συνδέονται με την ασφάλεια τροφίμων, όπως είναι και η υγεία των ζώων και των φυτών. Ε, κάνουμε επιστημονικές ε, γνωμοδοτήσεις για σας, τους νομοθέτες και ε, για εκείνους που διαχειρίζονται το κίνδυνο έτσι ώστε να βασίζονται οι αποφάσεις στην επιστημονική ε, συμβουλή που δίνουμε εμείς. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι δεν είμαστε ούτε ελεγκτές, ούτε αστυνομία, ούτε επιθεωρήσεις κάνουμε επιτόπου μας ζητούν επιστημονικές συμβουλές που βασίζονται σε δεδομένα και σε έρευνα. Και αυτό θέλει το χρόνο του και αυτό, για να συγκεντρώσει τα δεδομένα, να γίνει έρευνα κτλ. Ε, θα πρέπει ε, να τα κάνουμε όλα σωστά και εγκαίρως. Βεβαίως, Εργαζόμαστε με ταχύς ρυθμούς, αλλά η ποιότητα της παροχής συμβουλών εξαρτάται από την ποιότητα των δεδομένων που λαμβάνουμε και ε, συνήθως αυτά δεν έρχονται και ακαριέα. Χρειάζονται το χρόνο τους. Σας παραπέμπω στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων που είναι σε πολύ δινή θέση αυτή τη στιγμή γιατί θα πρέπει να εγκρίνει εμβόλια και χρειάζονται να έχουν τα σωστά δεδομένα πριν γνωμοδοτήσουν. Και εμείς λοιπόν πρέπει να έχουμε τα σωστά δεδομένα και την κρίσιμη μάζα των δεδομένων για να σας δώσουμε τη σωστή επιστημονική συμβουλή στην οποία θα βασίζετε τις αποφάσεις σας και τις μελλοντικές νομοθετικές σας ε, κινήσεις ε, από το 2002 λοιπόν έχουμε εκδώσει πάνω από 60 γνωμοδοτήσεις για την ευημερία των ζώων ε, από το 2004 μέχρι το 2010 είχαμε 58 γνωμοδοτήσεις, πολύ πύρετος. Μετά κάπως ηρέμησαν τα πνεύματα γιατί επικεντρωθήκαμε πλέον στην υλοποίηση της νομοθεσίας αυτής, στην εφαρμογή. Είχαμε άλλες 24 νομοδοτήσεις από το 2010 μέχρι το 2017 για διάφορα τέτοια θέματα. Και ε, χάρη και στις δικές σας πρωτοβουλίες πολύ πρόσφατα και τη καλή σας βοήθεια ε, έχουμε πάλι πολλή δουλειά ε, και περισσότερη για την ευημερία των ζώων και είναι σημαντικό να σας ευχαριστήσουμε. Το γνωρίζουμε ότι είναι χάρη σε εσά. Φυσικά εργαζόμαστε και για την υγεία των ζώων. Θα έχετε μάθει για την αφρικανική πανόλη του χείρου και πολύ πρόσφατα έχουμε τη γρήπη των πτηνών. Και μόλις τελειώσαμε την εργασία μας με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, ε, ελέγχου και πρόληψη νοσημάτων για τα βιζόν και τον κορονοϊό. Δηλαδή έχουμε δουλειά, δόξα τω Θεώ, και καλή συνεργασία. Ε, ας επικεντρωθώ τώρα σε αυτό που αφορά ιδιαίτερα τη δική σας Επιτροπή για τις μεταφορές των ζώων των ζώων. Έχουμε εκδώσει γνωμοδότηση το 2011 για τη μεταφορά των ζώων και με τη νέα στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο έχει εστιάσει εκεί ε, το ενδιαφέρον στην ευημερία των ζώων και έχουμε και επιπλέον εντολή, εντολές μάλιστα, όχι μόνο για τις μεταφορές των ζώων των ζώων, αλλά υπάρχει και μια ε, πρωτοβουλία ε, πολιτών για να τερματιστούν οι εκτροφές σε κλωβούς και για πτηνά ε, που εκτρέφονται για το κρέα τους, κρέας τους, για οτόκες όρνηθες ε, κλπ. Ε, υπάρχει και σαφής εντολή, πέντε εντολές είναι συνολικά, σαφή εντολή για τη μεταφορά των ζώων, την οποία έχουμε διαχωρίσει σε μεταφορά ζώων που εκτρέφονται ελεύθερα και ζώων που εκτρέφονται σε κλοβούς και είναι διαφορετικές οι γνωμοδοτήσεις που ε, θα βγουν. Έχουμε συστήσει ομάδες εργασίας που έχουν κάνει και τις πρώτες συνεδριάσεις και τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της συλλογή δεδομένων ε, και ε, συγκέντρωσης των επιστημονικών γνωμοδοτήσεων. Ας δούμε λοιπόν τις κατηγορίες που θα εξετάσουμε για κάθε μία από τις κατηγορίες ξεχωριστά. Ήδη μιλούμε για όλα τα ζώα που μεταφέρονται ζωντανά και για το καθένα από τα ζώα αυτά κοιτάμε τι γίνεται σήμερα, πώς μεταφέρονται, ποια είναι η πρακτική. Θα πρέπει να περιγράψουμε τι σημαίνει αυτό για την ευημερία τους, ποιοι είναι οι κίνδυνοι να τους ορίσουμε, να δίνουμε συστάσεις, έχουμε σαφή εντολή να σας δώσουμε και σε εσά και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή συστάσεις για να προλαμβάνονται, να ε, περιορίζονται και να διορθώνονται οι επιπτώσεις που έχουμε ε, εντοπίσει στην ευημερία των ζώων και ιδιαίτερα σενάρια κατά τη μεταφορά. Έχουμε πρακτικές δυσκολίες. Εσείς είστε σε καλή θέση, γιατί ήδη έχετε ακούσει την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ελεγκτικού Συνεδρίου και τη Γερμανική Προεδρία. Του Υπουργό Γεωργίας, που σας εξήγησαν ε, τι γίνεται και τι έλεγχοι έχουν γίνει. Και όλα αυτά τα λαμβάνουμε υπόψη και βλέπουμε τι προθυμία υπάρχει για να βελτιωθούν οι συνθήκες αυτές. Ε, θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Ε, ποιο είναι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Τελικά να έχουμε βελτιωμένες συνθήκες, όχι μόνο γενικότερα για την ευημερία των ζώων, και για την ευημερία τους κατά τη μεταφορά. Για τα σενάρια αυτά λοιπόν, όταν τα συζητούμε, θα πρέπει να συζητούμε και τι πρόκειται εμείς να κάνουμε. Ε, θα κάνουμε δημόσια διαβούλευση. Παρακαλώ, προσέξτε το. Στην αρχή Τη εντολής είχαμε σκεφτεί το Φεβρουάριο, αλλά μέχρι να στηθούν οι ομάδες εμπειρογνωμόνων χρειάστηκε χρόνος για να ρωτήσουμε ποια θα ε, μπορούσαν να είναι κάποια διαφορετικά σενάρια. Απαραίτητα, δεν ξέρω αν έχουμε παραλείψει τίποτα. Επίση, ζητήσαμε δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. και η δική σας Επιτροπή για τη Μεταφορά των Ζώων. Αν έχετε δεδομένα που δεν είναι ευρέως γνωστά και τα έχετε στη δική σας γνώση, παρακαλώ στείλτε τα και αυτά για να τα έχουμε και εμείς υπόψη μας. Προηγουμένως ανέφερα τον ΕΟΦ. Εδώ δεν μιλάμε για μαζικά δεδομένα δισεκατομμύρια ευρώ για φαρμακευτικές. Εδώ πρόκειται για ακτινιάτρους, ΜΚΟ, ανθρώπους που δουλεύουν στην πράξη, που έχουν δει κάποια δεδομένα, ορισμένα ερευνητικά κέντρα ε, στην ε, ε, πλατφόρμα, στα κέντρα αναφοράς. Αυτά τα δεδομένα συγκεντρώνουμε, αλλά δεν υπάρχει καμία μεγάλη βιομηχανία από πίσω. Είναι μάλλον μικρής κλίμακας και είναι δύσκολο να συγκεντρώσεις δεδομένα αλλά και πάρα πολύ κρίσιμο και σημαντικό. Και θα καλωσορίζαμε οποιαδήποτε στοιχεία θα μπορούσατε να μας δώσετε για να μας βοηθήσετε να προχωρήσουμε στην αποτίμησή μας και στην καλύτερη παροχή επιστημονικών συμβουλών. Νομίζω θα σταματήσω εδώ για να σας δώσω περισσότερο χρόνο σε εσά να κάνετε ερωτήσεις, να τοποθετηθείτε, να μας θέσετε υπόψη κάποια ζητήματα στην ΕΦΣΑ. Θυμηθείτε αυτό που είπε και η πρόεδρος, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Τώρα μόλις αρχίζουμε, τώρα πήραμε αυτές τις εντολές, έχουμε συγκεντρώσει τους εμπειρογνώμονες. Καμιά φορά δεν είναι και πολύ εύκολο, γιατί πολλοί από τους εμπειρογνώμονες έχουν, έχουν εργαστεί σε ΜΚΟ ή σε βιομηχανίες. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πάρα πολύ αυστηρή στη σύγκρουση συμφερόντων. Να έχουμε απόλυτη ανεξαρτησία στην παροχή επιστημονικών συμβουλών. Και θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ αυστηροί, επαναλαμβάνω, έτσι ώστε να είναι όλα ε, πεντακάθαρα, κρυστάλλινα και όχι επίμαχα. Ε, με χαρά θα συνεργαστούμε με όλους σας και θα ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι. Ευχαριστώ πολύ. Very much ε, for this Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτήν την ε, παρουσίαση. Με χαρά ακούσαμε ότι κάνετε πολύ σοβαρές αναλύσεις της κατάστασης και ναι, πρέπει να δώσετε μία σύσταση μέχρι τον Ιούνιο άνα είδος ε, ζώου για την μεταφορά των ε, ζών των ε, ζώων και βεβαίως νομίζω ότι όλοι μπορούμε με την ανταλλαγή των απόψεων να κάνουμε μια πολύ καλύτερη δουλειά. Οπότε, έχει τρία λεπτά ο καθένας. Ξεκινάμε με το ΕΛΚ και τον κύριο Ντανιέλ ε, Μπούντα. Έχετε τον λόγο για να κάνετε τις ερωτήσεις. Θα ακούσουμε πρώτα εσάς και μετά θα απαντήσει ο κύριος ε, Νικολάους ε, και ίσως και η Κομισιόν. Κύριε Μπούντα. Πατήστε το κουμπάκι παρακαλώ. Δεν σας ακούμε, το μικρόφωνο σας είναι κλειστό. Σας βλέπουμε, αλλά δεν σας ακούμε. Τώρα σας ακούμε. Θέλω να ευχαριστήσω τον προσκεκλημένο μας για τα όσα μας είπε. Εάν κατάλαβα καλά, είμαστε σε ένα στάδιο αξιολόγησης των προβλημάτων που υπάρχουν. Το έχω ήδη πει. Είμαστε σε ένα στάδιο αξιολόγησης, δηλαδή όσον αφορά την μεταχείριση των ζώων μέσα, ε, στις μεταφορές μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα έξω, προς τρίτες χώρες. Θέλω λοιπόν να σχολιάσω και να ρωτήσω το εξής. Πιστεύετε ότι οι εμπειρογνώμονες σας μπορούν να αξιολογήσουν την κατάσταση και σε τρίτες χώρες. Γιατί βέβαια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατά τη γνώμη μου, η κατάσταση είναι σχετικά απλή. Έχουμε την νομοθεσία, αποκτήσαμε και μία επιπλέον, γίνονται έλεγχοι στις διάφορες χώρες, αλλά μπορεί να υπάρχουν προβλήματα κυρίως όταν μιλάμε για εξαγωγές προς τρίτες χώρες. Γι' αυτό λοιπόν εδώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, σε τι βαθμό θα μπορούσε να γίνει μια αξιολόγηση της νομοθεσίας που ισχύει σε τρίτες χώρες. Τρίτες χώρες δηλαδή, αυτές με τις οποίες έχουμε ε, τέτοιου είδους ε, ανταλλαγές. Και να δούμε και κατά πόσο σέβονται την νομοθεσία και την καλή μεταχείριση των ζώων. Νομίζω ότι θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη μας και τα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών που έχουμε στην Ευρώπη. Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα με τους χείρους από την Κωνσταντσα. Στη συνέχεια εγκρίθηκε μια νομοθεσία στο Ρουμανικό Κοινοβούλιο, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις που κάνουν τις μεταφορές αυτές είναι υποχρεωμένοι να έχουν και δύο κτηνιάτρους καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς, οι οποίοι να μπορούν να διαβεβαιώσουν για την καλή μεταχείριση των ζώων μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, τέτοιου είδους παραδείγματα δεν θα έπρεπε να ισχύουν σε όλες τις χώρες μέλη. Ευχαριστώ. Thank you for these uh, two questions. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ε, δύο ερωτήσεις. Ε, δίνω τον λόγο στην κυρία Κάρμεν Αβραμ από τους σοσιαλιστές και δημοκράτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και σας κύριε Κρίς. Ο κανονισμός αυτός λοιπόν του 2005 μας παρέχει ένα πλαίσιο για την προστασία των ζώων κατά την μεταφορά όμως ε, η εμπειρία μας δείχνει ότι υπάρχουν δυσκολίες στην πρακτική εφαρμογή, δεν υπάρχει ομοιόμορφη ε, εφαρμογή, αποδεκτή θερμοκρασία, ελάχιστη χρόνη ταξιδίου και κυρίως υποτίθεται ότι θα είχατε ενημερωμένες λεπτομέρειες ανά είδος μέχρι τον Ιούνιο φέτος και κόβεται το σήμα. Η σύνδεσή μας ε, δεν είναι καλή. Θα προσπαθήσουμε να ξανασυνδεθούμε με την κυρία Αβραάμ. You can press the speak button, please. Πιέσατε το κομβίον, παρακαλώ. Αυτή είναι η κάμερα από την πίσω μεριά. Μπορείτε να αλλάξετε, σας παρακαλώ. Τώρα με βλέπετε. Ωραιότατα. Με ακούτε. Ναι, σας ακούμε, σας βλέπουμε. Όλα καλά. Ναι. Είναι κρίμα λοιπόν ότι η δική εκθέση δεν θα έρθει εγκαίρως για την δική μας, για να συντάξουμε την δική μας, αλλά όπως είπε ο κύριος Μπούντα εντωμεταξύ, κάποια κράτη-μέλη όπως η Ρουμανία ήδη προσπαθούσαν να βελτιώσουν ακριβώς ε, την ευσοία των ζώων και τη σχετική νομοθεσία. Οπότε, θα κάνετε κάποια βήματα για να ε, συστήσετε κάποια βήματα στους κτηνοτρόφου κατά τη διάρκεια των μεγάλων ταξιδιών και το τι πρέπει να γίνει με τα ζώα όταν φτάσουν στον προορισμό. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούσαμε τις ερωτήσεις. Ε, λοιπόν, Άσκαρ Κρίστενσεν τώρα από το Ρήνιο. Να το καλημέρα σας. Καλημέρα σας ε, και πάλι. Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο και ευχαριστώ και τον κύριο Κρίση για την παρουσίαση. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση αυτή για την ευζοία για κατά την μεταφορά και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον την έκθεσή σας ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια επικοδομητική συνεργασία. Για εμένα το θέμα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να υπάρχει, ε, υπάρχουν καλύτερες δυνατές ε, συνθήκες ε, για τα ζώα κατά την μεταφορά. Για μένα είναι εξίσου σημαντικό με τον χρόνο μεταφοράς των ζώων. Πριν από λίγα χρόνια ακολούθησα μία μεταφορά γουρουνιών από την Δανία στην Γερμανία. Εντυπωσιάστηκα από τις προσπάθειες οδηγών ε, αλλά και τους οδηγούς, κτηνοτρόφους και κτηνιάτρους που συνάντησα στη διαδρομή. Είμαι σίγουρος ότι κάνουν ό,τι μπορούν για να είναι άνετη η διαδρομή. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να γίνει αυτή ακόμα καλύτερα αν εκμεταλλευτούμε πλήρως τις τεχνολογικές να Έχω δει τα νέα φορτηγά που έχουν GPS, condition, συστήματα υπερήθρων, θερμομέτρησης και μέτρησης διοξιδίου του άνθρακα. Νομίζω ότι ε, αυτό θα οδηγήσει σε πολύ καλή ευζοία των ζώων και ταυτόχρονα θα διασφαλίσει ότι η υγεία ε, του ζώου θα είναι πολύ καλή κατά τη μεταφορά. Ε, θα έλεγα ότι θα ταξιδεύουν πρώτη θέση. Επίσης, η ΕΦΣΑ θα πρέπει να εξετάξει την δυνατότητα που δίνει η νέα τεχνολογία στον τομέα αυτών. Και δεύτερη ερώτηση. Έχετε κάνει κάποια μελέτη για το πώς σχετίζεται η φόρτωση και εκφόρτωση των ζώων με πιθανούς τραυματισμούς ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να συνεχίσουμε την συζήτηση. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας και θα δώσω τον λόγο στην κυρία Άνικα Μπρόνα, η οποία αντικαθιστά σήμερα την κυρία Λίμα από το ID. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Κρίτς στην μονάδα σας παραμβαίνετε και στις οζονώσεις. Κάτι πολύ σημαντικό, προκειμένου να έχουμε δεδομένα και να μας βοηθήσουν στην καλή μεταχείριση των ζώων. Μπορείτε να μας πείτε κατά πόσο η ΕΦΣΑ έχει εντοπίσει κινδύνους όσον αφορά την μεταφορά των ζώων όταν μεταφέρονται οδικώς αλλά και από τη θάλασσα. Υπάρχουν μέτρα έκτακτα στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια μόλυνση για να μπουν σε καραντίνα ή και για να τους προσφερθεί περίθαλψη. Ξέρουμε ότι τα κλωνοποιημένα ζώα κινδυνεύουν περισσότερο από τέτοιες μολύνσεις και κινδυνεύουν επίσης και να μεταδώσουν την μόλυνση εξαιτίας ακριβώς της γενετικής τους ιδιότητας. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε τη γνώμη σας για το... την κλωνοποίηση και τις οζωνώσεις, κατά πόσο δηλαδή η κλωνοποίηση ευνοεί την μετάδοση ε, των ασθενειών και μάλιστα προς τον άνθρωπο. Έπειτα η ΕΦΣΑ έχει πληροφορίες για μετάδοση του COVID-19 κατά την μεταφορά των ζώων. Προβλέπονται μέτρα για να αντιμετωπιστεί ένα τέτοιο δεχόμενο. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup pour ces questions. Σας ευχαριστώ. Η πέμπτη συντονίστρια είναι η Καρολίν Ροζ από τους Πράσινους. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ, κύριε Κρίτς, για την παρουσίασή σας. Η σύσταση που έγινε το 2011 από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων είναι πολύ διαφωτιστική, έχει επιστημονικά δεδομένα για να κρίνουμε ε, κατά πόσο υποφέρει κατά την μεταφορά ένα ζώο. Υπάρχουν οδηγίες ε, για το πώς θα φορτωθεί, για την μεταφορά, ανάλογα με τη μέθοδο μεταφοράς κτλ. Σε πολλά σημεία βλέπουμε ότι η επιστημονική γνώση θα έπρεπε να μας βοηθήσει να πάμε πιο μακριά από τον κανονισμό του 2005 όσον αφορά τους χρόνους μεταφοράς να είναι πιο σύντομοι, κυρίως για τα υποειδή, έπειτα ανάλογα ε, με το ζώο, ε, ο ύψος ανάλογα με το ζώο πάντα, ε, η θερμοκρασία πιο χαμηλή για τα πουλερικά κλπ. Και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν κέντρα υποδοχής, όχι μόνο για τα ζώα, αλλά και για τη δημόσια υγεία. Με τις ακροάσεις που κάναμε μέχρι τώρα φάνηκε ότι δεν εφαρμόζονται πάντα οι κανόνες. Και η δικιά σας έκθεση μας δείχνει ότι δεν φτάνουν μερικές φορές οι κανόνες. Οπότε πρέπει και να εφαρμόσετε καλύτερο κανονισμό του 2005, αλλά πρέπει και να ξαναγραφτεί. Μετά από αίτημα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, προχωρήσατε σε ενημέρωση των δεδομένων. Μας ε, μιλήσατε για πέντε εντολές και είπατε ότι μία διακριτή είναι αυτή για τη μεταφορά των ζώων. Αναφερθήκατε σε ζώα που εκτρέφονται ελεύθερα και άλλα που εκτρέφονται σε κλοβούς. Εγώ όμως θέλω να ρωτήσω πώς θα συμπεριλάβετε ή μάλλον θα συμπεριλάβετε στο έργο σας και θέματα τα οποία δεν αναφέρονται το 2011 την μεταφορά από θάλασσα, όταν μεταφέρονται τα ζώα δηλαδή ε, με πλοία για μέρες και μέρες προς τρίτες χώρες. Όταν ε, φορτώνονται στο πλοίο τα ζώα, τελειώνει ο έλεγχος. Δεν υπάρχει έλεγχος πια. Στην έκθεσή σας κάνετε κάποιες ε, διευκρινήσεις για τη θερμοκρασία, για το χώρο που πρέπει να έχει στη διάθεσή του το ζώο, αλλά Μερικέ φορές είναι τόσο συγκεκριμένε οι οδηγίες σας που αναρωτιέμαι μπορούν να ενσωματωθούν στο νόμο και θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και να ελεγχθούν. Στην έκθεση που ετοιμάζετε, τι θα κάνετε ώστε οι συστάσεις να εφαρμοστούν και να είναι εφαρμόσιμες πραγματικά για την καλή μεταχείριση των ζώων. Προβλέπετε λοιπόν να κάνετε γενικότερε συστάσει αλλά και συστάσεις οι οποίες να είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμε, να απαγορεύονται τα πιο μεγάλα ταξίδια, οι εξαγωγές ή η απαγόρευση μεταφοράς κάποιων συγκεκριμένων ειδών ζώων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ερωτήσεις. Τον λόγο έχει ο κύριος ε, Πέτερ Λοντγκρεν από το ECR. Καλημέρα. Καλημέρα συνάδελφοι. Την προηγούμενη εβδομάδα συναντήθηκα με τους Σουηδούς μεταφορείς ε, ζώων. Μία από τις πολύ δύσκολες καταστάσεις ε, που αντιμετωπίζουν είναι όταν έχουμε καύσωνα. Κάθε φορτηγό έχει ανεμιστήρες βεβαίως έτσι ώστε τα ζώα να έχουν μια ε, κανονική θερμοκρασία. Αλλά όταν υπάρχει καύσωνας, ε, η κατάσταση είναι δύσκολη. Καθώς μία ώρα πριν την άφηξη στο σφαγείο πρέπει να αναπαυθεί ο οδηγός για 45 λεπτά. Και όταν σταματάει ένα τέτοιο φορτηγό γεμάτο γουρούνια, για 45 λεπτά, τότε ε, όσους ανεμιστήρες και να έχει ε, δεν επαρκούν. Οπότε, εδώ οι οδηγοί έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα. Τι κάνουν. Θα παραβιάσουν τους κανόνες ε, ανάπαυσης ε, ή θα αναπαυθούν και όταν φτάσουν τελικά στο σφαγείο θα έχουν μερικά νεκρά ζώα και αυτό είναι επίσης ε, πρόβλημα και για τον οδηγό. Οπότε βεβαίω είχαν πρόβλημα γιατί ό,τι και να κάνουν θα τιμωρηθούν. Είτε θα παραβιάσουν τον χρόνο οδήγησης ε, είτε θα τιμωρηθούν επειδή θα φτάσουν με νεκρά ζώα και λυπούμε ε, γι' αυτό που θα πω αλλά δεν ε, έχουμε πολλά ντόπια σφαγεία πλέον. Στο όνομα του κέρδους ε, και του ανταγωνισμού η αγορά των σφαγείων έχει ε, γίνει πιο συγκεντρωμένη σε μεγάλα σφαγεία. Άρα θα υπάρχουν μεταφορές ε, που θα χρειαστούν κάποιο χρόνο. Δυστυχώς έτσι έχει η αγορά για να ε, υπάρχει κερδοφορία. Οπότε, το ερώτημά μου εδώ θα είναι το εξής. Τι κάνουμε για να διασφαλίσουμε ότι δεν θα τιμωρούνται οι οδηγοί, στο παράδειγμα που μόλις σας έδωσα. Τι κάνουν. Ε, συνεχίζουν να οδηγούν γιατί ο αέρας όταν κινείται το φορτηγό ε, κρατάει τη θερμοκρασία χαμηλή. Όταν σταματήσει λοιπόν το φορτηγό έχουμε πρόβλημα. Τι μπορούμε να κάνουμε ε, για να υπάρχουν πιο ευέλικτοι κανόνες για τους οδηγούς. Εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερο να συνεχίσουν να οδηγούν για άλλη μία ώρα από το να πεθάνουν κάποια ζώα στο δρόμο. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για να γίνει αυτό. Και επίσης θα ήθελα να γνωρίζω ποιες ε, είναι οι απόψεις για τις εναλλακτικές στρατηγικές όπως οικονομικότερα ή κινητά σφαγεία για κοντά στα αγροκτήματα, για άμεση πώληση που θα αντικαθιστούν την μεταφορά ζών των ζώων έτσι ώστε να μεταφέρονται μόνο σφάγια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις ερωτήσεις τελευταία ερώτηση από την κυρία Άνια Χάζεκαμπ από την Γκουε. Σας ευχαριστώ Τίλη, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε και εσείς κύριε Κλής. Πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια ζώα μεταφέρονται στην Ευρώπη σε μεγάλες αποστάσεις κάθε χρόνο. Και χάρη στο δικό μας ε, το σύστημα επικρατεί το οικονομικό συμφέρον και βρισκόμαστε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν έχει την υποχρέωση να το αλλάξει αυτό, να σταματήσουν να υποφέρουν τα ζώα κάθε μέρα στις ε, Μεταφορέ μεγάλων αποστάσεων. Είναι απαράδεκτο επί σειρά ετών οι ευρωπαϊκοί κανόνες να παραβιάζονται ε, διαρθρωτικά θα έλεγα όπω έχω παρατηρήσει και η ίδια. Οι κανόνες προφανώς δεν επαρκούν ε, για να προστατεύσουν τα ζώα κατά τη μεταφορά. Η αξιολόγηση της, του σχετικού κανονισμού μαζί με την αξιολόγηση του άλλου κανονισμού που αφορά την ευσογεία των ζώων είναι κάτι το οποίο πραγματικά απαιτείται επιγόντως. Είμαι απογοητευμένη για το ότι η προηγούμενη Κομισιόν σπατάλησε τόσο χρόνο ε, χρόνο κατά τον οποίο τα ζώα συνέχισαν να υποφέρουν. Δυστυχώς τώρα η Κομισιόν θα χρειαστεί άλλα δύο χρόνια για να κάνει αξιολόγηση. Ενώ το 2011, πριν από 10 χρόνια σχεδόν, η ΕΦΣΑ είχε ήδη καταλήξει πως ε, οι ε, μεταφορές μεγάλων αποστάσεων ε, είναι καταστροφή και αυξάνεται ο κίνδυνος ζωονόσων. Λοιπόν, εγώ θα εστιάσω τώρα στο δεύτερο συμπέρασμα της έκθεσής σας. Εάν μετά το 2020 δεν είναι ακόμα σαφές για το γιατί μπορούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην έχουμε ε, στο μέλλον ζωονόσους, ε, δηλαδή δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Έχουμε εδώ πέρα μια ορολογιακή βόμβα. Έχουμε τους ανθρώπους κλεισμένους στο σπίτι, αλλά τα ζώα μεταφέρονται από την Ολλανδία στην Κίνα και στη Ρωσία. Αγελάδες από τη Λιθουανία στο Ισραήλ και στο Λίβανο, πρόβατα από τη Ρουμανία στο Κουβέιτ, ε, αγελάδες από την Ιρλανδία στην Αίγυπτο κτλ. Και ενώ βρισκόμαστε εν το μέσο μιας τεράστιας κρίσης, μας περιμένουν και άλλες. Πριν από λίγες εβδομάδες υπήρχε μια, ένα νέο κρούσμα ε, πυρετού των χείρων στον Καναδά. Και στη χώρα μου, στην Ολλανδία, έχουμε πολλές ε, ζωονόσους. Από το 2007 πάνω από 130 άνθρωποι έχουν πεθάνει από ανθρωποζωονόσους και ε, διάφοροι άλλοι έχουν χρόνιες ασθένειες έχουμε γρήπη των πτηνών και αυτό το μήνα πάλι είχαμε μια τέτοια επιδημία και πάνω από 100 αγροκτήματα έχουν μολυνθεί με COVID και μιλάμε για ανθρώπους και γάτες και σκύλους. Κύριε Κρίς, εσείς ασχολείστε με την πανόλη των χείρων και βεβαίως ε, είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε τα αισθήματα. Οπότε η ερωτήση μου είναι η εξής πώς αντιδράτε όταν μία μελέτη της ΕΦΣΑ με τα συμπεράσματά της βρίσκεται στα συρτάρια της Κομισιόν επί 10 χρόνια χωρίς να αλλάζει τίποτα, όπως έγινε με την έκθεσή σας για τις μεταφορές μεγάλων αποστάσεων. Και αν οι μεταφορές είναι μία από τις πιο σημαντικές διαδικασίες διάδοσης ζωονόσων που μπορεί να γίνουν άνθρωπο ζωονόση. Συμφωνείτε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να σταματήσει αυτό, παραδείγματο χάρη, αλλάζοντα το αγροτικό μα σύστημα προ την τοπική και μικρή κλίμακα παραγωγή, μειώνοντα δραστικά το χρόνο μεταφορά χωρί καμία εξαίρεση όπως ε, γίνεται τώρα για τον χρόνο μεταφορών 8 ε, ωρών και άρα θα πρέπει να απαγορευτεί η εξαγωγή ζών των ζώων άπαξ και διαπαντός. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Άγια. Για τις ερωτήσεις θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Νικόλαος Κρίτς από την ΕΦΣΑ για 10 λεπτά για να απαντήσει σε όλες αυτές τις τόσο ενδιαφέρουσες ερωτήσεις πρέπει να πω. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τα μέλη της Επιτροπής. Όντως πολύ ενδιαφέρουσες, απαιτητικέ ε, και ποικίλε ερωτήσεις θα κάνω ό,τι μπορώ για να τις ε, διατρέξω από την αρχή μέχρι το τέλος και να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις ε, με όσο γίνεται αυτή τη στιγμή περισσότερες λεπτομέρειες. Θα επανέλθω στις πρώτες ερωτήσεις. Ο αξιότιμος κύριος Μπούντα ερώτησε για τις εξαγωγές, συμφωνίες, ευθέρωσης συναλλαγών και αξιολόγηση της νομοθεσίας. Ας απασχολεί αυτό και μας εμείς δεν μπορούμε να αξιολογήσουμε την νομοθεσία. Ούτε μέσα στην Ένωση, ούτε εκτός της Ένωσης. Εμάς επιστημονική γνωμοδότηση μας ζητούν για τις συνθήκες και συμβουλές, για το πώς μπορούμε να τις βελτιώσουμε. Αν θέλετε να το τραβήξω ε, και μέχρι την ερώτηση της κυρίας Χάζεπα, ε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Φυσικά να κάνουμε. Αλλά δεν χρειάζεστε την εύσα για να κάνετε ό,τι μπορείτε. Εμείς θα σας δώσουμε τα επιστημονικά στοιχεία. Το 2011 είναι πολλά χρόνια πριν. Είχαμε κάνει και τότε συστάσεις, θα τις ενημερώσουμε, υπό το φως των νέων γνώσεων, της έρευνας και των δεδομένων, των επιστημονικών. Αλλά, αν θέλετε εσείς να δράσετε, δεν χρειάζεται να μας περιμένετε εμάς. Εμείς συμβουλές δίνουμε και ε, εκτίμηση κινδύνου για να σας δώσουμε την ε, απαραίτητη επιστημονική αρρωγή, όπως λέει και ο τίτλος μας. Εμείς δεν μπαίνουμε σε συμφωνίες ελευθέρων συναλλαγών, ούτε σε νομοθεσία, ε, πόσο μάλλον εξωτερική. Αλλά μπορούμε να στέλνουμε και δύο κτηνιάτρους ε, στα πλοία βεβαίως και μπορεί να γίνει αυτό, η Ρουμανία το κάνει. Ή, ή άλλο εκπαιδευμένο προσωπικό, φυσικά. Αυτό είναι μουσική στα αυτιά μου, γιατί βελτιώνει την ευημερία των ζώων. Ε, Miss Ε, μετά, ε, για την επιστημονική γνώση και τα δεδομένα. Ε, για τις μεγάλες αποστάσεις, τα μακρινά ταξίδια, νομίζω σε αυτό απάντησα, για την νομοθεσία. Ε, είπατε για, την, για το συνοστισμό, για τον εξαερισμό, το μικροκλίμα ε, θα το κοιτάξουμε. Απολύτως, φυσικά, βεβαίως. Ε, θα τα ενημερώσουμε. Ναι, μιλήσατε για τις διακοιμάνσεις θερμοκρασίας κτλ. Ακριβώς αυτό είναι τμήμα της εντολής μας. Αυτό θα πρέπει να κοιτάξουμε, ε, να έχουμε όλα τα στοιχεία, να τα αξιολογήσουμε και μετά θα σας κάνουμε σαφείς συστάσεις. Έγινε και μια άλλη ερώτηση, νομίζω από την κυρία Ροζ, για το τι κάνουμε και πώς τα εφαρμόζουμε όλα αυτά. Προσπαθούμε να τα κάνουμε όσο γίνεται πιο εφαρμόσιμα. Αλλά από εκεί και πέρα η επιβολή και η εφαρμογή δεν είναι δικό μας θέμα. Είμαστε και πάρα πολύ μικρός οργανισμός, αλλά δεν είναι και στην εντολή μας. Δεν επιτρέπεται να κάνουμε κάτι τέτοιο. Κύριε Κρίστιανσεν. Για τις μεταφορές. όταν είναι πάρα πολύ υψηλής ποιότητας τα ζώα που μεταφέρονται ε, ε, θα πρέπει να φτάνουν σε όσο γίνεται καλύτερη κατάσταση εκεί που φτάνουν. Πολλές φορές είναι πολύ καλή η μεταφορά ε, και φροντίζουν πάρα πολύ, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις δεν ισχύει αυτό, το ξέρουμε. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το αρνούμαστε αυτό. Γιατί υπάρχουν ορισμένοι που παραβιάζουν ακόμα και την κείμενη νομοθεσία. Ε, νέε τεχνολογίε Ακούσατε τον Πέτερ Βέλτ από το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο και συμφωνώ και εγώ φοβούμαι. Ναι, η νέα τεχνολογία αν επιτρέπει να γίνεται καλύτερος έλεγχος, καλύτερη παρακολούθηση του μικροκλίματος που επικρατεί ε, στα μέσα μεταφοράς, ε, είναι και πολύ πιο φτηνή πλέον. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί βεβαίως. Εδώ η Amazon ελέγχει ε, τα δέματα που σας στέλνει και που βρίσκονται. Γιατί να μην μπορούν να ελέγχονται και τα ζώα που μεταφέρονται. Βεβαίως θα πρέπει εδώ να έχουμε υπόψη μας ε, θέματα προστασίας δεδομένων και θα τα κοιτάξει σίγουρα αυτά ο νομοθέτης με τις νομοθετικές του προτάσεις. Άλλο θέμα. Άλλη ερώτηση. Κορονοϊός και μεταφορές. με, την περασμένη Παρασκευή ε, εκδόθηκε ένα κείμενο που κάναμε μαζί με το ECDC ακριβώ για τα κράτη-μέλη για να φροντίσουν ε, για τη μεταφορά ιδίω των βυζών που είδαμε ότι ε, μεταδίδουν τον κορονοϊό και έτσι έχει συγκεντρωθεί η προσοχή και, και, και, μεταδότες και δεν συνιστάται προφανώς η μεταφορά βυζών αυτή την εποχή. Ευχαριστώ την κυρία Ρος. Συμφωνώ πολύ θα πρέπει να αναθεωρηθεί η νομοθεσία, να ξανακοιταχθεί, γιατί είναι το 2005. Βεβαίως, κάνετε κάναμε το 2011. για απαντώ και στην κυρία Χάζεκα εδώ. Για τα προσωπικά μου αισθήματα. Φυσικά θα πρέπει να εργαστούμε πιο σκληρά ε, έτσι ώστε η γνωμοδότηση του 2011 να ενημερωθεί καλύτερα. Είπαμε ήδη πόσο σημαντικό είναι να εργαστούμε για την ευημερία των ζώων. Και βέβαια σαφώς σήμερα βλέπουμε ότι ε, έχει γίνει και μόδα πολιτική. Εγώ δεν ε, καλούμε να αποφασίσω γιατί, αλλά να κάνω τη δουλειά μου γιατί είναι μια καλή ευκαιρία τώρα να κοιτάξουμε την ευημερία των ζώων, την μεταφορά τους και να την βελτιώσουμε περαιτέρω. Ε, γι' αυτό κάνουμε αυτή τη δουλειά και βρισκόμαστε εδώ που βρισκόμαστε. Καλά, τα ψάρια δεν είναι τμήμα της εντολής. Ειλικρινά δεν μας ζήτησε κανείς να κοιτάξουμε τι γίνεται με τα ψάρια. Είναι μεγάλες εντολές που έχουμε, και πέντε, και εκεί θα επικεντρωθούμε. Τα ψάρια εξαιρούνται. Αν καταφέρουμε ε, να ε, σεβαστούμε και το χρονικό πλαίσιο, θα είναι πραγματικά καλό το αποτέλεσμα, ελπίζω, για να βελτιωθεί η ευημερία των ζώων. Έχω και άλλες ερωτήσεις. Ε, εδώ σημειώσει ο κύριος Λούντγκρεν για τις μεταφορές στη Σουηδία. ανθρώπινη ευημερία απέναντι στην ευημερία των ζώων. Ο Ανδρέα Καβινέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε όταν έγινε ερώτηση στην τελευταία κρόαση. ότι είναι σε επαφή με τη Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και το κοιτάει και εμείς θα κάνουμε εκεί τις συστάσεις μας σίγουρα, αλλά οι νομοθέτες είναι εκείνοι που θα κάνουν τις νομοθετικές προτάσεις και να βρουν αυτή τη λεπτή ισορροπία. Όταν χρειάζεται πιο μακρά μεταφορά χρονικά ή όταν χρειάζεται να γίνονται τα διαλύματα ή παύσεις για ανάπαυση, ε, για να ποτιστούν τα ζώα κλπ. Το θέμα δεν είναι να γράφει κάποιες ρυθμίσεις σε ένα έγγραφο, αλλά να εφαρμόζεται με σαφή πληροφόρηση, να τα γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι, με φυλάδια, με υλικό. Γιατί οι περισσότεροι δεν θέλουν να παρανομούν, θέλουν να τηρούν τον νόμο, αλλά πρέπει και να τα γνωρίζουν με τρόπο εύληπτο. Επανέρχομαι τώρα στην κυρία Χάζεκαμπ. Δεν θα σχολιάσω ε, το τι συνέβη, δεν είναι ρόλος μου. Θέλω να επικεντρωθώ στη δουλειά που έχουμε εδώ και τι κάνουμε για την ευημερία των ζώων και καλύτερα αξιοποιώ το δικό μου και το δικό σας χρόνο. Τώρα που έχουμε την ευκαιρία μαζί σας. Να σας βοηθήσει αυτή η επιστημονική πλαισίωση ε, να νομοθετήσετε. Η αφρικανική πανόλη, θέλω να πω, δεν είναι ανθρωποζώο ε, έτσι μια μικρή παρατήρηση, γιατί ακούστηκε, δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο, δεν είναι ανθρωποζώο νόσος. Για τη μεταφορά των βυζών, σας είπα, μαζί με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων, το ECDC, κοιτάμε τις ανθρωποζωονόσους, ε, γιατί είναι γνωστές Και ε, αυτό οφείλεται στην εντατική γεωργία και κτηνοτροφία. Ούτε είναι μυστικό, δεν σας αποκαλύπτω τίποτα. Η εντατική ε, κτηνοτροφία οδηγεί και σε περισσότερους κινδύνους και ε, όταν παράγονται τρόφιμα από αυτά τα ζώα, τότε υπάρχει ένα θέμα ποιότητας, ποσότητας και ε, τιμής ε, της παραγωγής τροφίμων, που και αυτό είναι εκτό τη δικής μας εντολής. Εμείς θα πρέπει να σας δώσουμε τα επιστημονικά δεδομένα για να πάρετε εσείς αυτές τις αποφάσεις. Σταματώ εδώ, γιατί τελείωσε ο χρόνος μου και σίγουρα θα έρθουν και άλλες ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Thank you very much to you. Ευχαριστούμε πολύ. Όντως, απαντήσατε στις ερωτήσεις. Υπήρχε μια μικρή για την εξαγωγή σε ορισμένες χώρες. Στην αρχή ήταν αυτή η ερώτηση. Δεν σας άκουσα να αντιδράτε σε αυτό. Α, μιλήσατε λιγότερο από 10 λεπτά έτσι κι αλλιώς. Ίσως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει επίσης να απαντήσει. Οπότε αν έχουμε τον Κρίστιαν Ζούλιανσον από την Γενική Διεύθυνση Υγεία. Ίσως, αν θέλει, ευχαρίστω να προσθέσει και εκείνο τα δικά του σχόλια και απαντήσεις. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. αναφέρθηκε αναθεώρηση της νομοθεσίας μερικές φορές. Συμφωνώ. Η νομοθεσία του 2005 βασίζεται στην καλύτερη επιστημονική γλώση, γνώση που είχαμε τότε. Ε, προφανώς η ΕΦΣΑ σίγουρα θα συγκεντρώσει νέα επιστημονικά δεδομένα, διαθέτει νέα επιστημονικά δεδομένα με τα οποία μπορεί να αναθεωρήσει αυτή την νομοθετική ρύθμιση. Τώρα για τις τρίτες χώρες, τη διεθνή διάσταση για την οποία ρωτήσατε, ε, εθνική νομοθεσία και βέλτιστες πρακτικές. Όλα αυτά όντως θα ληφθούν υπόψη στο fitness check που κάνει τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα δούμε δηλαδή, όπως το έχουμε κάνει και παλιότερα, ποιες είναι μελλοντικέ ανάγκες. Όλα αυτά τα θέματα λοιπόν θα ληφθούν υπόψη και το θέμα των δικαιωμάτων των οδηγών για τον χρόνο ανάπαυσης, για παράδειγμα, σε σχέση με την καλή μεταχείριση των ζών. Ρωτήσατε ε, τι νόημα έχει να έχουμε για 10 χρόνια ένα καλό κείμενο στο γραφείο της Επιτροπής χωρίς να γίνεται τίποτα. Δεν είναι απόλυτα σωστό αυτό. Η έκθεση του 2011 της ΕΦΣΑ, που είναι η τελευταία επιστημονική γνωμοδότηση που διαθέτουμε για την ε, μεταφορά των ζώων από την ΕΦΣΑ, χρησιμοποιήθηκε, λήφθη υπόψη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της το 2011 για την εφαρμογή της νομοθεσίας του 2005. Και ναι, θα συμφωνήσω ότι υπήρξε κάποια διαφορά που εντοπίστηκε από την νομοθεσία και την υποστημενική γνώση. Κάτι το οποίο όμως αντιμετωπίστηκε με κατευθυντήριες γραμμές που προσθέθηκαν στην νομοθεσία. Επίσης εντοπίστηκε και ένα πρόβλημα που ακούστηκε και σήμερα και τις προηγούμενες φορές όσον αφορά την εφαρμογή ή το κατά πόσο είναι εφικτή η εφαρμογή της νομοθεσίας είναι και αυτή ε, μια δυσκολία με την οποία ασχοληθήκαμε πολλές φορές. Τα ακούσαμε και στις προηγούμενες συνεδριάσεις. Μιλήσαμε για πλατφόρμα που θα μπορεί να βοηθήσει τις διάφορες χώρες μέλη να ανταλλάσσουν ε, απόψεις, στοιχεία. Υπάρχουν πιλωτικά προγράμματα κλπ. κλπ. Ο κατάλογος είναι μακρύ Τώρα μπορεί κανείς να πει μα φτάνουν όλα αυτά ή δεν φτάνουν. Εντάξει, αυτά πάντως έγιναν στο παρελθόν. Μπορώ να ολοκληρώσω αναφερόμενοι στην απογοήτευση που αναφέρατε για το τι έκανε η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να ξέρετε ότι η Επιτροπή Βαντερ Λάιεν βάζει την καλή μεταχείριση των ζώων σαν προτεραιότητα. Και αν δείτε την επιστολή που έστειλε στην κυρία Κυριακίδη, αναφέρεται σε αυτά τα θέματα όσο επιτακτικά, όχι μόνο προτεραιότητα. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς θα φροντίσουμε να αναθεωρηθεί η νομοθεσία, η οποία θα βασιστεί βέβαια αναθεώρηση στα νέα επιστημονικά δεδομένα της ΕΦΣΑ και θα φροντίσουμε επίσης να μπορεί και εύκολα να τεθεί σε εφαρμογή. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Πράγματι, σας παίρνουμε κατά γράμμα με αυτά που είπατε, έτσι, ότι είναι όχι μόνο προτεραιότητα, αλλά και επιτακτικό για αυτήν την Επιτροπή. Θα δώσω τώρα το λόγο, ξεκινώντας το δεύτερο γύρο ερωτήσεων, στην Ελεονόρα Εύη. Μη εγγεγραμμένη. Δύο λεπτά παρακαλώ, Ελεονόρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον κύριο Κρίς ε, για την παρουσίασή του, την δουλειά που κάνει η ΕΦΣΑ είναι πολλοί τομείς ε, που αφορά αυτός ο κανονισμός για τη μεταφορά των ζώων και πολύ περισσότεροι ακριβώς ε, ε, οι διατάξεις εκείνες οι οποίες ίσως θα πρέπει να καταργηθούν. Θα ήθελα να αναφερθώ συγκεκριμένα σε ένα θέμα το οποίο αφορά την μεταφορά των ζώντων ζώων Συγκεκριμένα η ΕΦΣΑ είχε πει πως ε, δεν είναι δυνατόν πλέον τεχνικά τα ε, ζώντα ζώα να μεταφερθούν και την ίδια ώρα να ταϊστούν. Και βεβαίως γνωρίζουμε ότι οι ώρες ε, εκείνες οι οποίες διαρκούν ε, πάρα πολλέ ώρε. Παραδείγματο χάρη από την Ιρλανδία στην υπηρετική Ευρώπη, λαμβάνουν χώροι. Οπότε, αν ξέρουμε ότι δεν είναι δυνατόν τα ζώα να τα ειστούν κατά τη διάρκεια τη ε, μεταφορά, ε, θα έπρεπε ακριβώ να απαγορευτούν αυτά τα ταξίδια μεγάλη διάρκεια. Θα ήθελα λοιπόν εγώ να γνωρίζω τι γίνεται ακριβώς για τα ζώα εκείνα τα οποία δεν ε, τα ζώντα ζώα τα οποία είναι πέρα από την ε, μη ελάχιστη ηλικία κατά την οποία μπορούν τα ζώα να μεταφερθούν. Παραδείγματος χάρη όταν μιλάμε για μοσχαράκια τα οποία μεταφέρονται. Και τέλος ε, όσον αφορά τις ε, διαδικασίες ε, σφαγής ε, της ΕΦΣΑ όπου περιγράφονται στην έκθεσή σας οι κίνδυνοι που υπάρχουν για την ευζοία των ζώων και μιλήσατε για ανεπαρκείς αρμοδιότητες των αρχών. Τι γίνεται όμως με τις αρχές εκείνες οι οποίες ελέγχουν την μεταφορά των ζών Μήπως θα έπρεπε να έχουν περισσότερη βοήθεια και συγκεκριμένες δεξιότητες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσω τον λόγο στον Χουάν Ινάτσιο Ζόηρο από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ. Πριν διατυπώσω την ερώτησή μου, θέλω να ευχαριστήσω τους συντονιστές και την πρόεδρο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, ώστε να είμαι συνεισηγητής της έκθεσης που θα εκπονήσει η Επιτροπή μας. Ελπίζω να τα καταφέρω και να ανταποκριθώ στις προσδοκίες όλων όταν δημιουργήθηκε η Επιτροπή αυτή. Ο στόχος που έχουμε μπροστά μας είναι μεγάλος. Δεν πρέπει να προδώσουμε τις προοπτικές αυτές. Πριν να ασχοληθώ με την ε, πολιτική, ήμουν δικαστή στη χώρα μου και έτσι την εμπειρία μου θα ήθελα να την προσφέρω εδώ, ώστε να δούμε τι γίνεται με την ερμηνεία των διαφόρων νομοθετικών ρυθμίσεων με την συνεισηγήτριά μου και να καταλήξουμε σε ένα καλό αποτέλεσμα όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων. Γι' αυτό χρειαζόμαστε και τη συνεισφορά των συναδέρφων. Σήμερα ο κύριος Κρίτς έχει σίγουρα πολλά να μας πει. Περνάω λοιπόν τώρα στις ερωτήσεις μου. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Κρίτς για την παρουσίασή σας. Πιστεύω ότι ήταν διαφωτιστική. Θέλω να σας ρωτήσω για την κατάσταση όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάβασα στο βιογραφικό σας ότι έχετε περάσει από ερευνητικά πανεπιστήμια σε διάφορες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτός Ευρωπαϊκής Επίρου. Οπότε θέλω να μάθω κατά τη γνώμη σας. Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές μεταφοράς των ζώων ή που να είναι πιο απαιτητικέ από ότι είμαστε εμείς στην Ευρώπη. Μπορείτε να μου πείτε εάν υπάρχει κάτι που γίνεται κάπου αλλού στον κόσμο που εμείς θα έπρεπε να το αντιγράψουμε και πώς ή αντίθετα πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στην πρώτη γραμμή παγκοσμίω όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων κατά τη μεταφορά. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε μία νομοθεσία που θα έπρεπε να τη γράψουν άλλες χώρες αν όντω είναι έτσι, είναι πολύ σημαντικό. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υπάρχει μέσα σε ένα κενό. Όταν υπάρχει ζήτηση, όπου υπάρχει σήμερα από τρίτε χώρες για ζώα, ε, και θα πρέπει να γίνεται η μεταφορά. Και αν αντί για τη μεταφορά από την Ευρώπη, τα ζώα αυτά μεταφέρονται από άλλες χώρες, εκτός Ευρώπης, με λιγότερες απαιτήσει από αυτές που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν κάνουμε, δεν βοηθάμε τα ζώα έτσι. Όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, με τη διαρροή άνθρακα, αν περιορίσουμε την εξαγωγή ζώων από την Ευρώπη, κινδυνεύουμε να δημιουργήσουμε και μειωμένες προδιαγραφές όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων στη μεταφορά δεν είναι μόνο για να έχουμε η συνείδηση, είναι για να βελτιώσουμε πραγματικά την καλή μεταχείριση των ζώων. Γιατί αυτός είναι ο κύριος σκοπός μας εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Ευχαριστούμε πολύ. Χαίρομαι που σας βλέπουμε εδώ, που είσαστε συνεισήγητης. Η κυρία Ισαμπέλα Καρβάλης από τους Σοσιαλδημοκράτες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα. Καλημέρα, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Κρίτς για την σημερινή του παρουσίαση. Θέλω επίσης να τον ευχαριστήσω και για την ανεξαρτησία της ΕΦΣΑ όσον αφορά το έργο της ε, σε αυτό το τομέα που εξετάζουμε. Υπάρχει ένα θέμα που παραμένει από το 2011, το οποίο ήδη αναφέρθηκε τότε. Δηλαδή, οι περιορισμοί στη θερμοκρασία, οι βέλτιστες συνθήκες μεταφοράς. Θα ήθελα λοιπόν να ξέρω εσείς πώς βλέπετε ε, τις εξελίξεις από το 2011 και τι πρέπει να κάνουμε τώρα για αυτό το θέμα που είναι προτεραιότητα, ο εξαιρισμός κλπ. Ήδη από το 2011 είχαν ε, εντοπιστεί τα προβλήματα όσον αφορά τη θαλάσσια μεταφορά ε, ζώων. Υπήρχε μεγάλη μεγάλο ποσοστό θανάτων κατά τη μεταφορά αυτή εξαιτία ε, της αγωνίας που αντιμετώπιζαν τα ζώα κατά τη μεταφορά αυτή. Αυτό υπάρχει βέβαια και στις διεθνείς μεταφορές. Θα ήθελα να ξέρω, υπάρχει κάποια στρατηγική για τον εξαιρισμό που να είναι αποτελεσματική αλλά και ρεαλιστική και η οποία να επιτρέπει αποδεκτές συνθήκες για τα ζώα, τα οποία υποφέρουν από τις υψηλές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους. Ξέρω ότι η εντολή σας είναι απαιτητική, αλλά είναι και αναγκαία. Χρειαζόμαστε πολλά αξιόπιστα δεδομένα που να βασίζονται στην επιστήμη. Έτσι θα μπορέσουμε και εμείς να καθορίσουμε την ε, τοποθέτησή μας τελικά. Ξέρω ότι εμείς πρέπει να έχουμε τη δικιά μας έκθεση έτοιμη πριν από τη δικιά σας, οπότε δεν μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε, αλλά τουλάχιστον πείτε μας τη γνώμη σας για αυτά τα διάφορα ζητήματα που τίθενται όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων και που κατά τη γνώμη σας απαιτούν ακόμα περισσότερες έρευνες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Μάλεν Μόχτλοκ, ΕΛΚ, παρακαλώ τώρα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αξιότιμη κύριε Κρίς, εγώ είμαι από τη Βαβαρία. Τα δύο τρίτα του πλούτου της παραγωγής στη Βαβαρία είναι από την κτηνοτροφία. Γι' αυτό ε, γι αυτός είναι και ο λόγος που ευτυχώς υπάρχουν ακόμα πολύ μικρές ε, οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Γι' αυτό χρειαζόμαστε λύσεις και συστάσεις που να εξασφαλίζουν την επιβίωση αυτών των εκμεταλλεύσεων. Ερωτώ τα μοσχάρια γάλακτος πρέπει να τρώνε γάλα. Ε, στις μεταφορές έχουν άλλες προδιαγραφές από όταν μεταφέρονται ε, βόδια ε, ή μεγαλύτερη ηλικία μοσχάρια. Τι γίνεται με τους μόσχους γάλακτος. προτίθεστε να εξασφαλίσετε τη σωστή διατροφή τους. Έχετε λύσεις. Και τι γίνεται με την πραγματογνωμοσύνη και την εκπαίδευση, όχι μόνο για αυτά τα μοσχάρια γάλακτος, αλλά γενικότερα ε, για τα ζώα που μεταφέρονται. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές, για τα μοσχάρια που θυλάζουν ακόμα. Ο κύριος Μάρτιν ε, Χόισι από το ε, Ρινιού. Καλημέρα Μάρτιν. Καλημέρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ κύριε Κρίς και σας πρόεδρε, κύριος Χόισικ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση και χαίρομαι που συνεργάζεστε με την Επιτροπή μας. Πριν πω στην ερώτησή μου, έχω μια παρατήρηση, ένα σχόλιο που νομίζω ότι έχει σημασία. Νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι ότι η μεταφορά ζώων των ζώων είναι κάτι το οποίο στρεσάρει τα ζώα και η διάρκεια του ταξιδιού όπως και οι συνθήκες επηρεάζουν τα ζώα. Μιλάμε συνέχεια για το τι να κάνουμε, πώς να τα βελτιώσουμε όλα αυτά. Ε, εγώ έχω μια ερώτηση. Προσπαθούμε να ρυθμίσουμε και κάτι άλλο νομοθετικά. Δηλαδή να μην ενθαρρύνουμε έμεσα ή άμεσα ε, αυτά τα μακρινά ταξίδια ε, ε, ειδικά προσφαγή. Αφού πηγαίνουν στο σφαγείο έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορούμε να φέρουμε κοντά τα σφαγεία στην εκτροφή. Δεν μπορούμε να έχουμε περιφερειακά σφαγεία, ακόμα και τη σφαγή να υποστηρίζουμε στην εκτροφή. Αυτό δεν είναι μόνο καλύτερο για την ευημερία των ζώων, αλλά και για την ανάπτυξη της περιφέρειας και ε, τις μικρές εκμεταλλεύσεις και γενικότερα την ανάπτυξη της υπαίθρου. Έρχομαι λίγο στα επιστημονικά και συγγνώμη που μακρηγορώ. Θέλω να ρωτήσω τι θα γίνει με την επιστημονική γνωμοδότηση που θα εκδώσετε ε, ε, για τα ζώα. Συχνά τα πτηνά, τα κοτόπουλα και τα κουνέλια ε, τα παραβλέπουμε και ουσιαστικά τα μεταφέρουν σε κλουβιά, σε, σε κάτι κυβότια κοντέινερ θα τα χαρακτήριζα κιόλας. Ξέρουμε αυτό πόσο επιβλαβές είναι όταν μεταφέρουμε τα ζώα σε κλωβούς, όχι μόνο στα πουλερικά, και πηγαίνουν στα σφαγεία ε, παραμένοντας μέσα σε αυτά τα κλωβιά. Δεν θέλω να επαναλάβω κάτι που είπε μια συνάδελφος, αλλά γίνονται έλεγχοι σε όλα τα κρατη Μπορείτε να μας πείτε περισσότερα για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Ε, ε, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας και για όλο το έργο σας στην ΕΦΣΑ για να μας υποστηρίξετε και να μας βοηθήσετε ε, στη λήψη των αποφάσεων. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις αυτές, Μάρτιν. Ο κύριος Μοχάμεντ Σαΐμ, Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, τελευταίος ομιλητής για σήμερα. Καλημέρα σας. Κύριε Σαΐμ, ανοίξτε το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ε, ζητώ συγγνώμη. Νομίζω ότι ήταν ανοιχτό το μικρόφωνο. Καταρχά θέλω να σα ευχαριστήσω, Πρόεδρε, ε, ε, και εσά, κύριε Κρίση, για την παρουσίασή σα. Είναι σημαντική εντολή που έχετε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε πολλή δουλειά τα επόμενα χρόνια και εμεί για τη νέα νομοθεσία και μεταξύ ε, σημαντικών άλλων θεμάτων είναι και η μεταφορά. Εμείς δεν είμαστε ελεγκτές μέσα, είπατε, και επιθεωρητές. Ούτε εμεί. Αλλά αυτό που μα ενδιαφέρει είναι εφαρμόζεται η νομοθεσία, η κείμενη και η μελλοντική. Η καλή νομοθεσία είναι το πρώτο βήμα. Αλλά αν δεν μπορούμε να πιάσουμε τους κακοποιούς που την παραβιάσουν, δεν γίνεται τίποτα, δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό είναι θέμα των εθνικών αρχών και οργανισμών, αλλά στο παρελθόν έχουμε δει ε, ότι δεν ε, λειτουργούν όλα εύρυθμα σε όλα τα κράτη-μέλη. Ελπίζω η ΕΦΣΑ να βοηθήσει. Το ξέρω ότι εσείς κοιτάτε τα επιστημονικά και όχι την εφαρμογή, αλλά μήπως να συντονίζατε αυτή την εφαρμογή. Και αν όχι η ΕΦΣΑ, τότε κατά την επιστημονική σας άποψη ποιος θα πρέπει να επιληφθεί για την εφαρμογή του νόμου. Με ποιο τρόπο θα κάνετε μια προσέγγιση ειδική ε, προς το είδος του κάθε ζώου. Γιατί στο παρελθόν δεν υπήρχε αυτό και ήταν πολλά τα προβλήματα. Πώς θα τα λάβετε υπόψη όλα αυτά. Τελευταία ερώτηση και τελειώνω. Μιλήσατε για δεδομένα, αν έχετε στοιχεία δώστε τα. Μπορείτε να μας πείτε λίγο περισσότερο. Τι στοιχεία θέλετε να σας δώσουμε. Ποια είναι τα στοιχεία που σας λείπουν. Τι είδους στοιχεία δηλαδή ε, θα θέλατε να σας δώσουμε που υπάρχει έλλειμμα για να φροντίσουμε να το καλύψουμε αν μπορούμε. Θα ήταν πολύ χρήσιμο κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ για τις ερωτήσεις αυτές. Και τώρα και πάλι ο κύριος Κρίς, Δέκα λεπτά, αν και ξεπεράσουμε ήδη το χρόνο μας, 10 λεπτά για να απαντήσετε σε αυτές τις ερωτήσεις. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ελπίζω να με ακούτε καλά. Πρώτα απ' όλα ζητώ συγγνώμη για την παράληψη αυτή που επισημάνατε για τις εξαγωγές και τις συνθήκες της εξαγωγές που νομίζω αφορά και άλλες ερωτήσεις που έκανε ο κ. Ε, Τσόιντο και η κυρία Καβαλέ. Οπότε να αναφερθώ και σε αυτό αμέσως. Είναι μέρος της εντολής μας να κοιτάμε τους χρόνους και τις συνθήκες μεταφοράς και πέρα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε θα το δούμε αυτό. Βεβαίως ε, το τι σημαίνει αυτό νομοθετικά ε, επαφίεται σε εσάς, αλλά θα το εξετάσουμε γιατί αναφέρθηκε ήδη οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τα μεγάλα ταξίδια είναι ένα ζήτημα. Τώρα, δράτω με επίσης της ευκαιρίας να πω ότι ε, ε, κύριος Τζούλιαντσεν από την ε, Κομισιόν είπε κάτι το πάρα πολύ σωστό και δεν θέλω να δώσω λάθος εντυπώσεις γιατί πράγματι μετά από τη γνωμοδότησή μας η Κομισιόν εργάστηκε πάρα πολύ σκληρά στην εφαρμογή και νομίζω ότι η Κομισιόν αποφάσισε ότι το έχουμε ε, δει αυτό το εκμεταλλεύτηκε στο μέτρο του δυνατού και τώρα πρέπει να επανελεγχθεί ακριβώς για να δούμε πώς μπορεί να γίνει η νομοθεσία κατάλληλη για τον σκοπό της. Οπότε συμφωνώ πλήρως με αυτό. Τώρα, συγκεκριμένα για τις ερωτήσεις που αφορούν το ότι ο τρέχον κανονισμός δεν επαρκεί και το τι πρέπει να κάνουμε σχετικά. Κοιτάξτε, αυτό σχετίζεται και με την εφαρμογή σαφώς, αλλά α, προφανώς η Κομισιόν έχει κάνει αυτή την αξιολόγηση και έχει εξετάσει την σχετική αναγκαιότητα και θεωρεί ότι απαιτείται αναδιατύπωση, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει μια βελτίωση, ώστε αξίζει να το δούμε όμως. Πρέπει να πω και από την τελευταία μας γνωμοδότηση το 2011 κάποιες από τις συστάσεις που κάναμε τότε θα τις επανεξετάσουμε αλλά ίσως είναι οι ίδιες και ίσως ε, καταλήξουν στην νομοθεσία ή όχι. Αναλόγως βεβαίως και με τις ε, τεχνικές ε, λεπτομέρειες που θα θέλετε να μπουν στην νομοθεσία. Όσον αφορά τα γουρούνια, τα μοσχάρια που δεν έχουν απογαλακτιστεί είναι ένα συγκεκριμένο σενάριο που μας ζητήθηκε να εξετάσουμε και ζητώ συγγνώμη ακόμα δεν είναι δυνατόν να πούμε ε, το τι συστάσεις θα κάνουμε γιατί δεν είναι το τι θα πω εγώ αλλά η ειδικοί μας ε, μαζί με το πάνελ ευζοίας των ζώων ε, θα αξιολογήσουν και μετά ε, θα κάνουν τις ε, συστάσεις τους. Οπότε να περιμένετε νέα μας, αλλά δεν είναι κάτι στο οποίο μπορώ να απαντήσω τώρα. Ευχαριστώ κύριο Τσόιντο τώρα για τις δικές σας τις παρατηρήσεις. Θέλω να πω δύο πράγματα. Ναι, υπάρχουν άλλες χώρες, υπάρχει νομοθεσία σε άλλες χώρες. Έχω εργαστεί και στην Αυστραλία και στη ΣΥΠΑ και στην Ασία. Και οπωσδήποτε στην ε, Αυστραλία υπάρχει μια τεράστια συζήτηση για τη μεταφορά ζών των ζώων στη Μέση Ανατολή και οπωσδήποτε του απασχολεί το θέμα και γίνεται η ίδια συζήτηση αν πρέπει να απαγορευτεί. Αλλά η συζήτηση και η απόφαση αυτή είναι θέμα του νομοθέτη. Αυτό το οποίο μπορούμε εμείς να κάνουμε είναι να είμαστε σε επαφή με τον Παγκόσμιο Οργανισμό για την Υγεία των Ζώων και τον ΦΑΟ του ΟΗΕ για να ε, τους ενημερώνουμε και να τους δώσουμε την ευκαιρία να ευθυγραμμιστούν αν θέλουν, αλλά προφανώς η ΕΦΣΑ ε, δεν έχει νομοθετική αρμοδιότητα στην Ευρώπη και οπωσδήποτε δεν έχει εκτός Ευρώπης. Αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να σας δώσουμε τις επιστημονικές πληροφορίες. Ε, τώρα στην κυρία Καρβαλέ. Και πάλι εδώ μιλήσαμε για το τμήμα της εντολής, δηλαδή όρια θερμοκρασίας, ε, ταξιδιού, αερισμός. Σας διαβεβαιώ ότι αυτό είναι μέρος της εντολής μας, ε, ειδικά οι μικροκλιματικές συνθήκες. Ε, κυρία Μότλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, και εγώ είμαι από το Steiermark στην Αυστρία. Ε, το ξέρετε, έχει ακόμα πιο μικρές ε, ε, πιο μικρές εκμεταλλεύσεις. Ε, οπωσδήποτε υπάρχουν οι ίδιες δυσκολίες και ακριβώς σημασία των συστάσεων που αφορούν και τις μεγάλες μεταφορές είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μετά η ερώτηση για τα περιφερειακά σφαγεία το έχουμε συζητήσει, θα το ξανασυζητήσουμε. Το έχω δει και ως κτηνίατρος που έχω εργαστεί σε σφαγεία στο παρελθόν. Για να... Δηλαδή αν δείτε πώς έχουν μειωθεί, έχουν γίνει με, μεγάλα κεντρικά και τώρα τι πρόβλημα δημιουργεί αυτό με τον COVID. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές, ε, αλλά δεν είναι κομμάτι της εντολής μας βεβαίως, ότι εδώ ε, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά το τι μπορεί να γίνει καλύτερα με το επιπλέον όφελος στις μεταφορές βεβαίω που μπορεί να έχει. Μία ολιστική άποψη λοιπόν εδώ θα είναι υποφελής. Δεν αναφέρθηκα στις αρμοδιότητες γιατί είναι κομμάτι της εκπαίδευσης που έκανε και η Κομισιόν τα τελευταία χρόνια. Αφορά την συμμόρφωση και το πόσο, ε, σε ποιο βαθμό πάμε. Πάντα βεβαίως μπορούμε να κάνουμε κάτι ακριβώς για να βελτιώσουμε τα επίπεδα των δεξιοτήτων στα σφαγεία που είναι μεγάλο ζήτημα. Είναι ζήτημα κατάρτισης ε, ε, μισθών και οπωσδήποτε μπορούν να γίνουν βελτιώσεις σε σχέση με το συγκεκριμένο ερώτημα του κ. Χόισιν για τα χρόνους ταξιδιού σε κοντέινερ και τα λοιπά, τα είπαμε αυτά το 2011 και είπαμε ότι θα πρέπει να είναι τμήμα του χρόνου ταξιδιού έτσι ώστε συγκεκριμένα να ληφθεί υπόψη αυτός ο χρόνος ε, σκλοβούς ε, το εδώ τη σημειώση μου για την εφαρμογή. Ναι, δεν είναι ε, δική μας ε, δουλειά. Α, τώρα, ε, οπωσδήποτε, μια προσέγγιση αναείδος, ναι. Είναι κάτι το οποίο θα αναπτύξουμε και βεβαίως όσον αφορά το κενό των δεδομένων, εάν μου επιτρέπετε, παραδείγματο χάρη για την ιδανική θερμοκρασία για το κάθε είδος, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να έχουμε περισσότερα δεδομένα για την έρευνα. Ποια είναι η ιδανική θερμοκρασία, πώς αισθάνονται άνετα, χωρίς να υφίστανται ταλαιπωρία. Είναι ελάχιστα αυτά τα δεδομένα. Χρειαζόμαστε περισσότερα λοιπόν για τις συνθήκες μεταφοράς, τη διάρκεια της μεταφοράς, ένα ζήτημα οικονομικών συνθήκων ε, τα τελευταία δέκα χρόνια σημαίνει ότι δεν έχουμε την έρευνα που θα θέλαμε και θα σκοπεύσουμε με τον περιορισμένο προπολογισμό μας να δούμε συγκεκριμένες πτυχές αυτού του θέματος αλλά δεν είμαστε ερευνητικό ίδρυμα που μπορεί να χρηματοδοτήσει έρευνα αλλά εντός του προπολογισμού μας θα κάνουμε ό,τι μπορούμε έτσι ώστε να στοχεύσουμε και εμείς συγκεκριμένα κάποιες από τις ελλείψεις δεδομένων. Νομίζω απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Αλλά είμαι στην διάθεσή σας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε λεπτά ακόμα. Αν θέλει να αντιδράσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν λέω ότι είναι απαραίτητο, αλλά αν θέλει ευχαρίστω να ακούσουμε την Επιτροπή. Ο κύριος Γιούλισον. Αναφερθήκατε στην συμμόρφωση Εκεί είπατε ότι είναι στοιχείο κλειδί. Και η Επιτροπός Κυριακίδης, αλλά και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το 2012 αναφερόταν ότι προτεραιότητα δίνουμε στη συμμόρφωση. Η συμμόρφωση στους κανόνες λοιπόν είναι ευθύνη των χωρών μελών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει ό,τι μπορεί για να ελέγξει ότι γίνεται αυτή η συμμόρφωση από την Γενική Διεύθυνση που τώρα είναι η ΣΑΝΤΕ και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και στο μέλλον η συμμόρφωση στους ισχύοντες κανόνους εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρόεδρο. ευχαριστούμε πολύ και περνάμε στον τρίτο γύρο ερωτήσεων από τους ευρωβουλευτέ. Ξεκινάμε από τη Χωσάνα Κόντε. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ και με συγχωρείτε δεν μπόρεσα να ακούσω όλους τους ε, παραμένοντες. Σας ευχαριστώ όμως για την παρουσίασή σας. Πράγματι υπάρχει ανάγκη ε, να αλλάξουμε τον κανονισμό του 2005. Δεν υπάρχει παγκοσμίω κάποια νομοθεσία πιο προχωρημένη για την μεταφορά των ε, ζώων. Έχουμε λοιπόν πάρα πολλούς κανόνες που επιβάλλονται στους μεταφορείς και τους ε, κτηνοτρόφους και κάνουν πολύ δύσκολη την δραστηριότητά τους. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Κρίντσι αν ε, μπορείτε να μας πείτε πού συγκεκριμένα δεν εφαρμόζονται ή παραβιάζονται πιο συχνά οι κανόνες και τι μπορεί να γίνει στην πλευρά των ελέγχων ε, στην κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το να απαγορεύσουμε τώρα τη μεταφορά ζών των ζώων στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι καταστροφικό για πολλού ε, τομεί ε, και για την ε, ζωοτεχνία, ειδικά στην ιστορική καμπή στην οποία ζούμε. Θα μπορούσαμε ίσως, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα, να μεταφερθεί Ίσως θα μπορούσαμε να απαγορεύσουμε την μεταφορά των ζώων προς τρίτες χώρες. Τι γίνεται λοιπόν. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα μπορούσαν να απαγορευτούν, εκτός βεβαίως από τις μεταφορές εκείνες στις οποίες πηγαίνουν για σφαγή για κάποιες θρησκευτικέ ανάγκες και τελετές. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε κάποιες εγγυήσει ότι τηρούνται οι δικέ μας οι Θα μπορούσαμε ίσως να έχουμε κάποιες διμερείς ε, συμφωνίες. Τώρα όσον αφορά την ευζοία των ζώων κατά την έκτροφη, ε, διάβασα τα έγγραφα τα οποία μας ε, δώσατε τα οποία ζήτησε η Επιτροπή μας, ε, δηλαδή ως επιστημονική γνωμοδότηση. Λοιπόν, έχουμε και τις ε, χερσαίες μεταφορές ε, τελικά. Αυτές είναι οι πιο μεγάλες και βεβαίως και οι θαλάσσιες, όπως είπαν και οι συνάδελφοι. Οι θαλάσσιες μεταφορές προς την Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ζώα ετησίως. Οπότε μπορούσε να γίνει ίσως μια μελέτη ad hoc ε, για τις ε, μεταφορές αυτές ε, προς το εξωτερικό εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, χερσαίες και θαλασσίες και θα ήθελα να μάθω τι σκοπεύει να κάνει η Κομισιόν και η δική σας υπηρεσία από αυτού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, Ευχαριστούμε και να τηρείτε το χρόνο σας παρακαλώ. Για τελειώς δεν θα μπορέσουν όλοι να πάρουν το λόγο και θα είναι κρίμα. Και φαίνεται υπήρχε πολύ αντίχηση και ήταν δύσκολο για τους διερμηνείς να σας μεταφράσουν. Τόμας Βάιτς τώρα από τους Πρασίνους. Παρακαλώ Τόμας. Καλημέρα σας ε, κύριε Κρές θα μιλήσω ε, κανονικά γερμανικά, τη διάλεκτο της Τυρίας δηλαδή, για να καταλαβαίνόμαστε και <laughs> να μεταφραζόμαστε. Ευχαριστώ για ε, την πρόσκληση να σας δώσουμε στοιχεία. Ε, είναι πιο φιλικό από αυτά που άκουσα από τον προϊστάμενό σας στην Επιτροπή που ασχολείται με τα φυτοφάρμακα. Θέλω να σας ρωτήσω έχετε κάνει μελέτες για την αντοχή ε, στα αντιβιωτικά, ε, ιδιαίτερα από περιοχές ε, που έρχονται τα ζώα, που έχουν πολύ εντατική κτηνοτροφία. Έχετε κάνει συστάσεις στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εφαρμοστούν για να βελτιωθεί η υγεία του πληθυσμού. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να σταματήσουν τελείως οι μεταφορές από ε, ε, αυτές τις περιοχές. Μιλήσατε για την Αφρικανική Πανόλη του Χείρου. Μήπως να απαγορευτούν τελείως οι μεταφορές ζών των χείρων. Τι λέει η Εύσα. Αυτά για τα δεδομένα. Ε, ε, ε ακραίες θερμοκρασίες. Έχετε στοιχεία για αυτές τις ακραίες θερμοκρασίες σε πλοία. Θα σας ήμουν ευγνώμων να μας τα δίνατε. Επίσης, σε όλα αυτά τα θέματα αναφέρομαι στη δική σας έκθεση του 2011. Έχετε στοιχεία για τα πλοία ότι ε, ε, επιτρέπεται πρόσβαση για ελέγχους και επιθεωρήσεις και υλοποιείται από αρμόδιες αρχές ε, είτε αυτή είναι κτηνίατρη είτε επίσημες αρχές επιθεωρήσεις. Έχετε στοιχεία και εμπειρίες επίσης Είπατε σε κάθε μακρύ ταξίδι και στα πλοία ε, να υπάρχει εκπαιδευμένο προσωπικό. Μπορεί να υπάρχουν ζώα εκεί ε, τραυματισμένα ή άρρωστα και θα πρέπει να θανατώνονται όπως πρέπει. Έχετε υπόψη σας ε, στοιχεία για τέτοιες περιπτώσεις ή δεν σας έχει απασχολήσει αυτό καθόλου. Και το τελευταίο για τα συστήματα εξαερισμού για να νεώνεται και να μπαίνει καθαρός αέρας και εκεί χωράει βελτίωση. Έχουν γίνει κάποιες βελτιώσεις. Έχετε στοιχεία συγκεκριμένα με ελέγχου τι γίνεται με τις θαλάσσιες μεταφορές προς τη Μέση Ανατολή. Να γίνεται σωστός εξαερισμός και σε περίπτωση που χαλάσει κάποια γεννήτρια. Και αν έχετε τέτοια στοιχεία θα μπορούσατε σας παρακαλώ να τα διαβάσετε στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ, Τόμας Φάιτς. Ιδιαίτερα, ναι, για τα στοιχεία και τα δεδομένα. Καλό είναι για εμάς γιατί είμαστε εξεταστική επιτροπή και είναι και τόσο ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Να μπορούσαμε να έχουμε και εμείς τα στοιχεία. Θα δώσω το λόγο πάλι στον Πίτερ Λούντκρεν από το ΙΣΙΑ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω και άλλες ερωτήσεις όταν πρόκειται για την αρμοδιότητα του οδηγού. Έχει κάποια πιστοποιητικά. Σημαίνει ότι είναι σε θέση να ασχοληθούν με τα ζώα. Και κανονικά οι επιχειρήσεις φροντίζουν, ξοδεύουν και χρήματα ώστε να έχει τα προσόντα που χρειάζεται ο οδηγός για να μπορεί να τα βγάλει πέρα σε μια κατάσταση αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα καταφέρνουμε αρκετά καλά. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια περίοδος κατάρτισης ε, πριν να αναλάβει μια διαδρομή μόνος του οδηγός. Δεν το έχουν αυτό όλοι. Το βλέπουμε και στους οδηγούς στην κυκλοφορία. Μερικές φορές αναρωτιέται κανείς για κάποιον άλλον οδηγό, μα πώς κατάφερε και πήρε δίπλωμα αυτός. Έτσι λοιπόν κάτι αντίστοιχο δεν θα έπρεπε να υπάρχει κατάρτιση για τους οδηγούς υποχρεωτικά και περίοδος άσκησης. Έπειτα δεν θα έπρεπε στην ίδια μεταφορά να είναι αρσενικά και θηλυκά. Ε, μπορεί να έχουν ζήσει μερικές φορές πολλά χρόνια μαζί και μετά η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη αν προσπαθήσει κανείς να χωρίσει τον αρσενικό τάβρο για παράδειγμα από τα θηλυκά. αν έχουν συνηθίσει να συνυπάρχουν, είναι πιο επικίνδυνο να προσπαθήσουμε να χωρίσουμε τα αρσενικά από τα θηλυκά και να τα μεταφέρουμε χωριστά. Ποια είναι η δικιά σας η γνώμη. Τι νομίζετε ότι θα μπορούσε να γίνει γι' αυτό. Ευχαριστούμε για αυτή την πολύ ιδιαίτερη ερώτηση. Τελευταία. Ο κύριος Παλάς Σιφέγγι από το ΕΛΚ τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι. Η υιοθέτηση της νομοθετικής ρύθμισης το 2005 έχει ξεπεραστεί βέβαια. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Τώρα, αυτοί που θέλουν να κάνουν πιο αυστηρό τον κανονισμό αυτό, δεν νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο περισσότερο πρέπει να επικεντρωθούμε στην συμμόρφωση που αναφέρει ο κανονισμός αυτός. Και να πούμε πού είναι τα προβλήματα με την συμμόρφωση. Η κατάρτιση είναι ένα θέμα. Ο χρόνος, η διάρκεια μεταφοράς κλπ. κλπ. Είναι πολύπλοκο βέβαια το θέμα και πολύπλευρο, αλλά έχει να κάνει κυρίως με τις εταιρείε μεταφοράς ζών. Θέλω να ρωτήσω πρώτον, ψηφιοποίηση. Κατά την επιστημονική σας άποψη, θα επικεντρωθείτε περισσότερο στις νέες τεχνολογίες και την χρήση τους, την ευρεία χρήση τους από πλευρά των εταιριών αυτών. Η Χούντλαντ, που είναι μια τέτοια εταιρεία στη χώρα μου, την Ουγγαρία, έχει μια νέα εφαρμογή που μπορεί και υπολογίζει το χώρο που έχει στη διάθεσή του το κάθε ζώο κατά τη μεταφορά. Είναι ένα παράδειγμα. Δεύτερον, δεύτερη ερώτηση η πρωτοβουλία για τους κλοβούς. Η παραγωγή όν στην Ουγγαρία αποφάσισαν για ενισχυμένους κλοβούς 100 εκατομμύρια ευρώ. Όταν κάνετε συστάσεις, θα λάβετε υπόψη σας και όλες τις περιπτώσεις τεχνολογίας που αφορούν τις οτόκες όρνηθες. Έτσι θα μπορούσε να υπάρχει μια πιο καλή βάση για να συγκρίνουμε τα διάφορα στοιχεία νέων τεχνολογιών και για τους ενισχυμένους ε, εμπλουτισμένους κλωβούς και για τη θερμοκρασία κτλ. Ό,τι αλλαγές πάντως γίνουν θα πρέπει να εξηγώνται ξεκάθαρα από τις μελέτες που γίνονται. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, Ευχαριστούμε. Ο τελευταίος τώρα σε αυτό το γύρο είναι ο κύριος Νίλ Σιμπουρξαμ, Σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ. Ο κύριος Φούλξ Ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ και την Εύσα που ήρθε για να συνομιλήσει μαζί μας. Με τον Έσκα που μίλησε νωρίτερα από το ΡΙΝΙΟΥ ήμασταν μαζί στην Επιτροπή για την μεταφορά των Ζών και συμφωνώ ότι οι προδιαγραφές που είδαμε εμείς ήταν πολύ καλές. Όμως φαντάζομαι ότι δεν εφαρμόζονται γενικά. Για παράδειγμα το όριο των 8 ώρων Σίγουρα χρειάζεται όριο στη διάρκεια. Αυτό βελτιώνει τη μεταχείριση των ζώων. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω την Εύσα να εξετάσει ή αν το έχει κάνει να μας πει ποια είναι η σχέση ανάμεσα στις γενικές συνθήκες καλής μεταχείρισης των ζώων και τις συνθήκες μεταφοράς τους. Η θερμοκρασία δηλαδή, η τροφή, το νερό, επαρκής χώρος κατά την Εύσα Υπάρχει σχέση ανάμεσα στις γενικές συνθήκε μεταφοράς και αυτές τις συγκεκριμένες παραμέτρους. Από τις πληροφορίες που έχω και από τους συνομιλητές μου φαίνεται πως υπάρχει σύνδεση. Δηλαδή ότι όσο μεγαλύτερης διάρκειας είναι η μεταφορά, τόσο πιο εύκολο είναι να παραβιαστούν αυτές οι παράμετροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ναι, Νίλς, θα ήθελα να το ξέρω, γιατί και εσύ και Σκαρ είπατε ότι βλέπετε καλές πρακτικές μεταφορές των ζώνων όταν ξέρανε δηλαδή οι μεταφορείς ότι εσείς θα πηγαίνατε ίσως. Νίκολας Κρίτσ τώρα και πάλι από την ΕΦΣΑ για να απαντήσει σε αυτόν τον γύρο ερωτήσεων. 10 λεπτά το πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ξεκινήσω από την πρώτη ερώτηση. Κυρία Κόντε, ευχαριστώ και για το σχόλιο για τις προδιαγραφές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ρωτάτε για τις υψηλές προδιαγραφές, εμένα για την Αυστρία, σαν να ρωτάτε την Αυστριακή ομάδα τι προδιαγραφές έχει. Πάντα μπορεί κανείς να τα καταφέρει καλύτερα και επαγγελματική μου άποψη είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση όντως έχει υψηλέ προδιαγραφές καλής μεταχείριση των ζώων, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε περισσότερα και να έχουμε ακόμα καλύτερες συνθήκες. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Μίλησαμε και πριν για μεταφορά ζών προς τρίτες χώρες και τις πληροφορίες που έχουμε. Εδώ επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ελεκτικό συνέδριο, το οποίο εκπώνησε έκθεση, πολύ καλή έκθεση, με στοιχεία από τις διάφορες χώρες. Δεν είναι δικιά μας εντολή να προβαίνουμε στους ελέγχους, αλλά όταν μας στάνουν πληροφορίες εννοείται ότι τις ελέγχουμε και τις λαμβάνουμε υπόψη. Το κύριο Βάτση θέλω πραγματικά να τον ευχαριστήσω. Γιατί ανέφερε αυτό ακριβώ που χρειάζεται, τα δεδομένα και γιατί εμείς κάνουμε δημόσια διαβούλευση, γιατί ακριβώς προσπαθούμε να εντοπίσουμε πού μας λείπουν στοιχεία και δεδομένα. Και εσείς κάνατε ένα πάρα πολύ ωραίο κατάλογο των δεδομένων τα οποία μας λείπουν. Όλα αυτά τα οποία παραθμίσατε πραγματικά είναι οι ελλείψεις μας. Προσπαθούμε να καλύψουμε αυτά τα κενά λοιπόν και γι' αυτό και έχουμε και τους εμπειρογνώμονές μας. Ζητώντας ε, αυτά τα δεδομένα, τη γνώση. Όταν δεν την έχουμε, φροντίζουμε να υπάρχει μια διαδικασία βάσει της οποίας την ζητάμε για να την έχουμε. Είναι μια μεθοδολογία που είναι πολύ αυστηρή ακριβώς για να εμποδίζουμε παρεκκλήσεις από τους κανόνες. Γι' αυτό και χρειάζεται χρόνος. Από την εμπειρία που έχουμε εδώ, αν πρέπει αυτό να γίνει online, χρειάζεται ακόμα περισσότερος χρόνος. Αλλά, εν πάση δικό μας είναι αυτό το πρόβλημα, δεν είναι δικό σας. Τώρα για το MR και τις μεταφορές. Η εντατική, δηλαδή, κτηνοτροφία. Υπάρχει έκθεση της ΕΦΣΑ, που έγινε σε συνεργασία μαζί μας από γιατρούς και άλλους ειδικού και είδαμε μεγάλη μείωση, κάτι το οποίο οδήγησε σε μείωση των αντιβιωτικών και μείωση τελικά της αντίστασης. Προσπαθώ εδώ τώρα να δω έχετε αναφερθεί σε διάφορα είδη μεταφοράς. Αυτό που θέλω να προσθέσω είναι ότι φυσικά και μπορεί κανείς να κάνει πολλά πράγματα στις μεταφορές των ζών. Ένα ακραίο παράδειγμα, ήμουνα και στη μεταφορά υποειδών, σε, με αεροπλάνο. Είναι θέμα φυσικά, τιμής και τα λοιπά, αλλά σήμερα πρέπει κανείς να έχει υπόψη του την τιμή και εμείς τονίζουμε και είμαι σίγουρο ότι και η Επιτροπή αλλά και εσείς θα φροντίσετε που μπαίνει το όριο. Γιατί εμείς βέβαια σας δίνουμε δεδομένα για την κατάσταση των ζών κατά τη μεταφορά, εσείς θα βάλετε το όριο τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι. Αυτό είναι προνόμιο και ευθύνη του νομοθέτη. Εμείς έχουμε την υποχρέωση να σας δίνουμε τα δεδομένα και τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Κύριε Χάνκτον, και εσείς θέσατε ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα για το αν πρέπει να χωρίζονται στις μεταφορές στάβρια από αγελάδες. Το 2011 δεν το αναφέραμε ρητά, αναφερθήκαμε στην ανάμειξη διαφορετικών κατηγοριών ζώων είναι κάτι που μπορούμε να εξετάσουμε. Και ακριβώ και εδώ πρέπει να συστήσουμε πού υπάρχουν ειδικέ περιπτώσεις. Μέρος της διαβούλευσής μας είναι ακριβώς και τέτοια πράγματα. Εσείς βάζετε τώρα ένα σενάριο εδώ δηλαδή το οποίο όντως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας για το χώρο, για τη θερμοκρασία, για τις μικροκλιματικές συνθήκες, για τον εξαιρισμό, πόσα τετραγωνικά ε, μέτρα ανά κιλό ή αν ότι όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία είχαμε θίξει το 2011 και θα τα επικαιροποιήσουμε εννοείται και τώρα. Δεν πρόκειται για το τέλος των ε, κλοβών αλλά σίγουρα δουλεύουμε και πάνω σε αυτό το θέμα. Ποιε είναι οι οικονομικές επιπτώσεις, όμως είναι εκτός της εντολή μα. Αυτό είναι κάτι το οποίο εσεί, οι νομοθέτες αποφασίζετε για το πόσο πολλά μπορούν να γίνουν έτσι ώστε και οικονομικά να είναι εφικτό κάτι, γιατί κανείς δεν θέλει να νομοθετήσει φυσικά σε ένα παράλληλο κόσμο. Προφανώ πρέπει να νομοθετήσει ο νομοθέτης κάτι το οποίο να είναι εφαρμόσιμο. Άρα εσεί θα αποφασίσετε για τι τιμές και τις αξίες. Τώρα είπατε ότι πήγατε σε μεταφορά ζών. 8 ώρες έχουμε πει ε, ότι είναι ένα σύντομο ταξίδι. Τώρα το σύντομο είναι σχετικό βέβαια. 11 είναι πολύ παραπάνω. Οι 30 ώρες εννοείται επιβάλλονται κανόνες εκεί και για παύσεις διακοπές λοιπά. Πρέπει να δούμε όντως πού πρέπει να υπάρχουν κτηνίατροι μαζί, που πρεπει να υπαρχουν εκτινίατροι μαζι που οχι Και έρχομαι και στις αρμοδιότητες των οδηγών. Δεν απάντησα σε αυτό. Και εδώ πολλά είναι εφικτά εφόσον υπάρχει πολιτική βούληση για την καλή μεταχείριση των ζώων, να εμπλέκονται κτηνίατροι. Εγώ στον καιρό μου το είδα να υπάρχουν ε, κτηνιατρικές ε, υπηρεσίες. Με τον αυτό διπηρετό μετά επίσης είδα πώς ε, υπήρξαν τελικά πολύ περισσότερο παντού. Αυτό είναι θετικό φυσικά για τους κτηνιάτρους και για όλους όσοι ασχολούνται με τα ζώα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες όντως θα έπρεπε να επανδρώνονται ικανοποιητικά και να έχουν τη δυνατότητα στις διάφορες χώρες να παρεμβαίνουν. Αυτό ξέρουν, αυτή είναι η δουλειά τους. Το ίδιο και για τους ελέγχους. Υπάρχουν διαφορές στους ελέγχους που γίνεται στις διάφορες χώρες. Μερικές φορές γιατί δεν υπάρχει αρκετό προσωπικό. Και υπάρχει και μια άλλη ερώτηση του κυρίου Βάιτς για τις μεταφορές σίγουρα ζώα τα οποία είναι μολυσμένα ασθενή με τον ένα τον τρόπο εννοείται ότι απαγορεύεται να ταξιδεύουν αυτό προβλέπεται ήδη όπου όμως η AFS δεν είναι παρούσα εκεί μπορεί να μην εφαρμόζεται αυτό. Να μην υπάρχουν τα σωστά μέτρα ελέγχου δηλαδή των ε, ασθενειών. Οι διάφορες παραβάσεις τώρα που γίνονται όσον αφορά τη θερμοκρασία, τον εξαιρισμό, νερό, πρόσβαση στο νερό, σε τροφή. Ναι, όσο πιο μεγάλης διάρκειας είναι το ταξίδι, όντως τόσο μεγαλύτερο είναι και ο κίνδυνος κάποια στιγμή να μην τηρούνται οι προδιαγραφές που πρέπει. Είναι ένας κίνδυνος ο οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί για να αντισταθμιστεί αυτό. Και αυτό θα κάνουμε. Και ό,τι άλλες ανησυχίες ή πληροφορίες έχετε, παρακαλώ να μας ενημερώνετε. Γιατί έτσι καλύπτεται τα δεδομένα που μας λείπουν. Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη αν μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Και πάμε στο τελευταίο γύρο των ομιλητών. Η κυρία Ζουλή Λεσαντέ. Euh, Ευχαριστώ, ε, Πρόεδρε ε, Κύριε Κρίτς, θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή σε μία έννοια που θα πρέπει να μας απασχολήσει. Είναι η αλυσίδα των ζωντανών οργανισμών και η διατροφική αλυσίδα υπάρχει ε, στο κρέας η αλυσίδα του ψύχου που θα, πρέπει να διακόπτεται με πολύ συγκεκριμένη χνηλάτιση και δρακόντιους ελέγχους για να είμαστε σίγουροι ότι αυτά τα ευπαθή προϊόντα ε, μεταφέρονται και στα ψυγεία, στα φορτηγά υπάρχει ένας μετρητής που μετράει το θερμόμετρο, ε, τη θερμοκρασία και αν για τεχνικούς λόγους, μηχανικούς ή λόγω αμέλειας ε, σταματάει το ψυγείο φαίνεται αυτό αμέσως στο μαύρο κουτί. Αυτό το μαύρο κουτί εξετάζεται λοιπόν συστηματικά κατά την άφηξη του φορτηγού πριν ξεφορτωθεί το εμπόρευμα δεν υπάρχει τίποτα σχετικό για τη μεταφορά ζών των ζώων και η χνηλασιμότητα ε, περιορίζεται στην ταυτότητα του, του ζώου με το ενότιο, ας πούμε, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα για τις συνθήκες μεταφοράς. Αν έχει ταϊστεί, αν έχει υποτιστεί σωστά ε, ε, και πώς έχουν γίνει όλα αυτά. Και υπάρχει και το θέμα του στρες, και, από το οποίο μπορεί και να ψοφήσουν τα ζώα. Σε περίπτωση, δηλαδή, ε, υπερκόπωσης και στρες φτάνουν στο σφαγείο άρρωστα τα ζώα. Γι' αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε αυτή την έννοια της αλυσίδας των έμβιων όντων, ε, γιατί έχει επιπτώσεις και στη δημόσια υγεία και στον άνθρωπο τελικά αυτό. Merci beaucoup pour Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις αυτές. Η Πρόεδρος θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Μανουέλα Γκρίπα των Πρασίνων Ελεύθερη Ευρωπαϊκή Συμμαχία. Γεια σου Μανουέλα. Ευχαριστώ ε, Τίλη. Αγαπητέ κύριε Κρίτς, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, στη στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο έχετε λάβει εντολή πολύ συγκεκριμένη. Η ΕΦΣΑ θα πρέπει να ενημερώνει με όλα τα στοιχεία για να μειώνεται ε, η επιβάρηση και η καταπώνηση των ζώων. Όλα αυτά είναι καλά νέα. περιμένουμε εδώ και καιρό αυτά τα δεδομένα. Πώς θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές και εμείς τι θα κάνουμε για να βελτιώσουμε την νομοθεσία. Στο παρελθόν έχουμε αποτύχει. Θα πρέπει η συστάσεις σας να είναι κάτι παραπάνω από ευχολόγια και ευσεβής πόθη. Και αυτό ε, δεν είναι μόνο δικό μας θέμα όπως υπενηχθήκατε, αλλά είναι και δικό σας θέμα. Η δική σας ε, υπηρεσία, η ΕΦΣΑ, πώς θα συνεργαστεί για να εφαρμοστούν αυτές οι νέες κατευθυντήριες γραμμές. Θα κάνετε σαφείς συστάσεις σε περίπτωση σοβαρών, επανειλημμένων κινδύνων και προβλέψιμων. Δεν μπορείτε να απαγορεύσετε, να βοηθήσετε να απαγορευτεί ε, ας πούμε η εξαγωγή τέτοιων ζώνη ή πολύ μακρινές ε, αποστάσεις που διανύονται. Είναι βάναυση αυτή η συμπεριφορά στα ζώα και μια προβοκατόρικη ερώτηση στο τέλος. Η καλύτερη σύσταση από πλευρά σας δεν θα ήταν να σταματήσουν τελείως ε, αυτά τα μακρινά ταξίδια και μεταφορές σε τόσο μακρινές αποστάσεις και να σπάζονται επιτόπου τα ζώα. Ευχαριστώ. Θα δώσω και πάλι το λόγο στην κυρία Νίκα Μπρούνα που το ξαναζήτησε. Ε, για να ξανακάνει τις ερωτήσεις της γιατί δεν απαντήθηκαν όλες για την κλωνοποίηση και κάτι άλλο. Ε, σας δίνω και πάλι το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περνάνε τα χρόνια, οι εκθέσεις, οι συζητήσεις, αλλά κάθε μέρα ε, ε, ε υποφέρουν τα ζώα στις μεταφορές γιατί παραβιάζονται οι κανόνες, η νομοθεσία δεν είναι αρκετή, χωρίς να αναφέρω ε, τις εξαγωγές προς χώρες Μαγκρέμπ και Μέσης Ανατολής όπου θανατώνονται βάναυσα και με πάρα πολύ ομό τρόπο. Ε, μήπως έχει έρθει η ώρα να επικεντρωθούμε ε, στη μεταφορά κρέατος, σφαγίων με γιώτα και όχι ζών των ζώων. Και αυτό απαντάει και στον κίνδυνο της σου και που τον εξαλείφει ουσιαστικά. Ε, αυτές είναι νέε ερωτήσεις και ζητώ συγγνώμη από τους διερμηνείς γιατί την η εικόνα. Θα δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Τόμας Βάιτ και πάλι των Πρασίνων για τις τελευταίες ερωτήσεις του πρωινού. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Κύριε Κρίς, σας ρώτησα από πού παίρνετε τα δεδομένα σας, από ποιους οργανισμούς ε, και πού βασίζετε την ενημέρωσή σας. Παρακαλώ μπορείτε να μας πείτε από πού αντλείτε αυτά τα στοιχεία. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο αν γίνεται στον κύριο Νικολάος Κρίς για πέντε λεπτά. Δεν θέλω να έχουμε υπέρβαση ωραρίου κάθε φορά. Αλλιώς οι διερμηνείς θα μας μποϊκοτάρουν. Thank you. Thank you very much. And I keep it short Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος ε, ε, γιατί σέβομαι πάρα πολύ τους διερμηνείς. Ε, το πρώτο, μεταφορά ζών των ζώων και πάλι έχουμε ένα σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που λέγεται traces και ειχνηλατεί ακριβώς τη μεταφορά. Υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Σε ό,τι αφορά τις συνθήκες, το μικρό κλίμα όπως περιγράψατε που επικρατεί, ε, υπάρχουν διάφορα μαύρα κουτιά που καταγράφουν αυτά τα δεδομένα. Φυσικά πάντα βελτιώνεται κατά κατάσταση, χωράει βελτιώσεις. ειδική αναφορά ε, στις μικροκλιματικές συνθήκες. Στη συνέχεια, η κυρία Ρίπα ρώτησε θα πρέπει να απαγορεύσουμε. Κοιτάξτε, δεν είμαι εγώ κατάλληλο για να σα πω, δεν είναι στη δική μα εντολή να σα πω τι ε, θέλω να απαγορευτεί. Και απάντηση να σα δώσω θα είναι προσωπική και όχι επαγγελματική από την ΕΦΣΑ και σίγουρα όχι ε, κάτι που βοηθάει να προαχθεί η συζήτηση. Αυτό έχει να κάνει με αρχές και ε, το τι είναι αποδεκτό και τι όχι. Ε, ε, δικό σας προνόμιο να τα λάβετε αυτά υπόψη. Εμείς σας λέμε τι σημαίνουν όλα αυτά για την ευζοία των ζώων. Ελπίζουμε να υπάρχει ένα μετρήσιμο επίπεδο. Ε, πώς ανεβαίνει η ευζοία και η ευημερία των ζώων. Ποια είναι ιδιαίτερα αρνητικά φαινόμενα. Και εσείς θα αποφασίσετε που υπάρχει το όριο του παραδεκτού και του απαράδεκτου. Το, αν θα απαγορευτεί κάτι ή όχι είναι στα χέρια του νομοθέτη, όχι της ΕΦΣΑ. Το αφήνω εδώ. Ε, κυρία Μπρούνα, για το κρέας. Και μεταφορά κρέατος σφαγίων ε, αντί για ζώντα ζώα. Ε, ναι, όταν έχουμε μόνο σφάγια που μεταφέρονται, δεν υπάρχουν τα ζητήματα που τίθενται με τη μεταφορά ζών των ζώων. Αλλά η απόφαση για το πώς θα πρέπει και πότε θα πρέπει να απαγορεύονται εντός ή εκτός της Ένωσης, οι μεταφορές ζών των ζώων. Αυτό σίγουρα θα είναι τμήμα της συζήτησης ε, και των θεμάτων που σας απασχολούν. Όπως σας είπα, η δική σας ε, αρχή είναι και δικό σας προνόμιο αυτό. Εμείς να σας βοηθήσουμε όπως μπορούμε. Γίνεται αυτή η συζήτηση, εμείς μπορούμε να σας δώσουμε επιστημονική βοήθεια ε, για τις συζητήσεις σας. Για τον κύριο Βάιτς, από πού αντλούμε τις πληροφορίες μας και τα δεδομένα. Από κέντρα αναφοράς, από πανεπιστήμια προσπαθούμε που εργάζονται για την ευζοία των ζώων, από τους επιχειρηματίες βέβαια που να μπορούμε να τα ελέγξουμε και να τα επαληθεύουμε και από διεθνή στοιχεία, κοιτάμε και τη βιβλιογραφία και μπορώ να το πω και με κάποια περηφάνεια ε, ότι διακρινόμαστε σε αυτό γιατί αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό κάνουμε συνέχεια. Και φυσικά θα τα δημοσιεύσουμε. Γνωρίζετε πολύ καλά ε, τι ισχύει για τη διαφάνεια και τι θα τεθεί σε ισχύ το Μάρτιο 2027. Όλα αυτά θα είναι στη διάθεση του κοινού και θα μπορείτε να τα ελέγξετε, να τα τσεκάρετε, να τα επαληθεύσετε, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν θέλουμε να κρύψουμε τίποτα. Ίσα ίσα. Αυτά αποτελούν τη βάση των συστάσεών μας. Ελπίζω να απάντησα. κοιτάμε διάφορες εκθέσεις, ε, βιβλιογραφία, δημοσιευμένη και μη. Ε, έχουμε ε, μια επισκόπηση όλου του πεδίου και βλέπουμε τι κυκλοφορεί. όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται στη γνωμοδότηση. Πολύ χρόνο σας έφεγα και ευχαριστώ και τους διερμηνείς και την Επιτροπή σας. Thank you very much uh, to you. Uh. Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κρίς για την παρουσίασή σας και τις απαντήσεις που δώσατε σε όλες τις ερωτήσεις και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον κύριο Κρίστιαν Τζούλιανσον, που απάντησε και εκείνο σε κάποιες ερωτήσεις. Σίγουρα καταλάβαμε ότι η ΕΦΣΑ γνωμοδοτεί, δίνει επιστημονική γνώση και συμβουλές, αλλά ε, πραγματικά ε, περιμένουμε από εσά πολύ ισχυρές συστάσεις. Εκεί έχετε ελευθερία και θέλω να ευχαριστήσω επίσης όλους τους συμμετέχοντες. Σήμερα το πρωί ήταν πολλοί κόσμος και πάρα πολλοί διαφορετικές ερωτήσεις. Ακόμα και αν δεν μπορέσαμε να μπούμε σε λεπτομέρειες στις απαντήσεις, νομίζω ότι ήταν πολλά τα σημαντικά θέματα που συζητήσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη συνεδρίαση. 2 Δεκεμβρίου. Και εκεί μπορώ να σας επιβεβαίωσω από τώρα ότι θα έρθει. Ο Επίτροπος Βοητσεχόφσκι, Επίτροπος Γεωργίας, ε, ελάτε κι εσείς, προσέχετε μέχρι τότε και τα λέμε. Γεια σας.